Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα μάθατε ότι χθε ε, σε ένα αυτοκινητόδρομο της Γερμανίας έλαβε χώρα ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα με ένα λεωφορείο με Πολωνούς τουρίστες ε, που προερχόταν από την Ισπανία και χτυπήθηκε, συγκρούστηκε με μια ιδιωτική χρήση Mercedes χρειάστηκε να βγει από το δρόμο και χτύπησε σε μια γέφυρα το λεωφορείο. 13 ε, έχασαν τη ζωή του ε, και κάποιες δεκάδε είναι τραυματισμένοι, μερικοί σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Θα ήθελα να σα ζητήσω να κρατήσουμε ενό λεπτού σιγή για τα θύματα αυτού του τραγικού τροχαίου που έλαβε χώρα χθε στη Γερμανία. Okay, thank you, Mrs. Asadi. Yes, can we just stand then for a moment, please? Λοιπόν, αν θέλετε να σηκωθούμε όλοι, ε, να τηρήσουμε ένα λεπτού σιγή για τα θύματα αυτού του τροχαίου δυστυχήματος. Dziękuję bardzo. E, thank Dziękuję bardzo. Okay, ladies and gentlemen, you have before you the uh, draft. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχετε το σχέδιο ημερησίας διάταξης, έχετε κάποιο σχόλιο. Ναι, υπήρξαν κάποιες αλλαγές, αλλά αυτό γιατί προσπαθήσαμε να δούμε τι μπορεί να γίνει με το πρόγραμμα αν συμφωνείτε, στη συνέχεια έχουμε την έκδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων, αφού εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αξιολόγηση τη προοδού εξέταση των υπολογιών. Κυρία Μάισνερ, έχετε το λόγο. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Bei dem Bericht Σα ευχαριστώ. Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ε, η βασική μου ε, ανησυχία ε, και βασικό μου μέλημα ήταν να λάβω υπόψη αυτά τα οποία έχουν λεχθεί μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, έχουμε τη γαλάζια βίβλο, έχουμε τα πράγματα τα οποία ήδη έχουν εφαρμοστεί, αυτά τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν για να ε, εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτή την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρξουν επικαλύψεις ε, και ε, θα ήθελα να σας πω ότι εμένα με απασχολεί κυρίως η διακυβέρνηση, η επιτήρηση και ο στόχος είναι να ε, βρούμε κάποια κοινά διαβήματα. 104 τροπολογίες υποβλήθηκαν. Θέλετε να περιμένω λίγο. Τι θέλετε, Πρόεδρε, να συνεχίσω, γιατί... Να. 104 τροπολογίες, λοιπόν, ε, και γενικά πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι ε, οι ομάδες συμφώνησαν και χαίρομαι ιδιαίτερα. Βεβαίω πρέπει να συνεχίσουμε την επεξεργασία αυτή τη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, να την εμβαθύνουμε και φυσικά ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μερικέ φορέ τα στοιχεία ε, θα διαφέρουν μεταξύ του, αλλά άλλε φορέ θα οδεύουν προ την ίδια κατεύθυνση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιου συμβασμού και θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτού του συμβασμού. Εσεί στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκα με του κοιόδου ηγητέ. Συζητήσαμε σε βάθο το ζήτημα και νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ε, ευρεία συμφωνία. Ε, ο κατάλογος είναι διέτοιμο, παρόλο που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε σε ορισμένα σημεία ε, κάποια στοιχεία, γιατί κατατέθησαν τις άλλε τροπολογίες. Και βεβαίω, όσον αφορά τις προφορικές τροπολογίες, ε, θα αναφέρω ε, τη δική μου θέση. Για να εξετάσουμε του συμβιβασμού Πρώτα απ' όλα τον Α. Πρόκειται για, θαλάσσιες θαλάσσια παράδοση, για την θαλάσσια ανάπτυξη. Όλες οι μελέτες που έχουμε σχετικά με τις ε, προβλέψεις για το μέλλον προβλέπουν σημαντική ανάπτυξη των παρακτήων περιοχών. Έτσι λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητο και σκόπιμο να προωθήσουμε αυτήν την διάσταση της πολιτικής 2020. Έχουμε καταλήξει σε ένα συμβασμό που νομίζω ότι θα ικανοποιήσει τους πάντες. Τώρα, συμβασμός Β. Εδώ μιλούμε για την οικολογική καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού. Το έγραφα εγώ στην εκθεσή μου αυτό, τα σχετικά δηλαδή, αλλά όλοι βέβαια κάθισαν και σκέφτηκαν πώς μπορεί να γίνει καταπολέμηση τέτοιων ε, φαινομένων στο μέλλον με καλύτερο τρόπο και να αποφευθούν κυρίως, να προληφθούν οι καταστροφές αυτές. Και αυτές οι τροπολογίες λοιπόν κατέληξαν σε ένα συμβιβασμό των υπαριθμών Β. Ο Γ βεβαίως μιλεί για ολοκληρωμένη πολιτική θαλάσσης που θα χρειαστεί, αν θέλει να αναπτυχθεί, και ειδική χρηματοδότηση. Και εδώ έχουν γίνει διάφορες προτάσεις που συγχωνεύσαμε σε ένα συμβασμό Γ. Αυτές οι, αυτοί οι συμβασμοί ήταν σχετικά απλή. Δεν ήταν βέβαια όλοι απλοί. Ο Δέλτα που έχει ε, σχέση με την ε, εποπτεία των θαλασσίων περιοχών εκεί υπήρχαν διαφορές απόψεων. Συζητήσαμε διαμακρών, καταλήξαμε ωστόσο σε συμβαστική πρόταση που νομίζω ότι θα ικανοποιήσει την πλειοψηφία. Διότι αφενός χρειαζόμαστε έλεγχο, χρειαζόμαστε εποπτεία, αλλά δεν θέλουμε να είναι υπερβολικά αυτά. Ούτε θέλουμε να ε, χειραγωγούμε εμεί τι χώρες μέλη σε αυτές τις δράσει. Ο συμβασμό ε, η αρχική μου παράγραφος 28, είναι αυτή που έδωσε αφορμή σε περισσότερε συζητήσεις αλλά και κάποιε παρανοήσει. Εγώ είχα γράψει στην έκθεσή μου πρόγραμμα ανανέωση στόλων. Δεν εννοούσα βέβαια ότι οι πλουσιότερες χώρες θα πρέπει να χρηματοδοτούν τις για να αγοράσουν καινούργια σκάφη. Στην ε τώρα πάντως που έχουμε καταθέσει είναι πιο ξεκάθαρο το νόημα. Δηλαδή ότι εδώ στην ε, Ευρώπη έχουμε πολύ τεχνογνωσία σχετικά με το λεγόμενο green shipping Βρισκόμαστε λοιπόν πολύ μπροστά, έχουμε σημαντική πρωτοπορία και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη τεχνογνωσία ώστε να αναλάβουμε ένα ρόλο ηγετικό ανά τον κόσμο. Αυτό εννοούμε στην ε, συμβαστική τροπολογία ε. Τώρα η σίγμα ταφ, η F, που είναι και η τελευταία, αναφέρεται στον τουρισμό. Ο τουρισμός εντάσσεται και αυτός στην ολοκληρωμένη πολιτική της θάλασσας. Και ειδικά ο τουρισμός σε ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές πρέπει να γίνεται με τρόπο αηφόρο, βιώσιμο, γιατί έχει βέβαια σχέση και με την αυσιπλοεία και με κάποια επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν έχουμε πάλι συμπεριλάβει τις διάφορες τροπολογίες. Αυτά σχετικά με τις τροπολογίες συμβιβασμού. Αυτό που θα ήθελα τώρα να ακούσω, τι έχουν να πούν οι σκιώδεις συζητητές δηλαδή σχετικά με την πρόοδο των συζητήσεων, χθε αλλά και σήμερα νομίζω κατατέθηκαν από το Λαϊκό Κόμμα ορισμένες προφορικές τροπολογίες. Με τον σκιώδη συγητή κ. Κουμουτσάκο συζητήσαμε και διμερό, διότι υπήρχαν πολλές τροπολογίες οι οποίες κάπως μου φάνηκαν ε, πολύ μακροσκελεί. Δηλαδή επί της ουσίας ναι μεν μπορούσα να τις υποστηρίξω, αλλά δεν ήθελα η έκθεση να γίνει τόσο μεγάλη. Ήθελα λοιπόν να εξετάσω μαζί του πώς μπορούμε κάνοντας συντομότερες διατυπώσεις, να γίνει και πιο σφιχτή η έκθεση, να μην είναι βαρετή στο διάβασμα, στο πω έτσι. Λοιπόν, καταλήξαμε σε κάποιες κοινέ τροπολογίες, τις οποίες θα υποστηρίξω σε μεγάλο βαθμό. Θέλετε να σας πω ποιες προφορικές θα υποστηρίξω και ποιες όχι. Κύριε Αντιπρόεδρε. Όχι. Καλώς. Καλά λοιπόν αυτές, αυτά σχετικά με τις νέες. Ε, Α, ναι. Μια στιγμή όμως πρέπει να πω κάτι ακόμη. Τροπολογία 27. Θα την υποστηρίξω, αντιθέτως από αυτό που αναγράφει η λίστα ψηφοφορίας. Σημαντικό λοιπόν να σας το πω αυτό. «25 το πρώτο μέρος όχι». Τώρα οι προφορικές μια στιγμή να βρω το έγγραφο, οι προφορικές τροπολογίες που κατατέθηκαν τώρα, αφενός η 9, θα την υποστηρίξω, 39 του Λαϊκού Κόμματος. Αυτές είναι του Λαϊκού Κόμματος. Θα την υποστηρίξω επίσης. 45, επίσης νέα αυτή. Α, όχι, όχι, όχι, όχι, υπήρχε ήδη από πριν. 51 την υποστηρίζω. 52 όχι, δεν θα την υποστηρίξω, διότι εκεί πάει να γίνει μια επικάλυψη και δεν έχω καμία αντίρρηση για την Union of the Mediterranean, δεν έχω καμία αντίρρηση να αναφερθεί, αλλά έχει αναφερθεί και αλλού και τότε θα έπρεπε να περιλάβουμε και άλλες μακροστρατηγικές περιφέρειες. Επίσης, 55 και εδώ προβλέπεται προφορική τροπολογία την οποία δεν θα μπορέσω να υποστηρίξω πάλι από το ΕΛΚ 84 και 88 μαζί επίσης δεν μπορώ να υποστηρίξω διότι έχουμε άλλες τροπολογίες, άλλες διατυπώσεις 97 και 98 θα υποστηρίξω καθώς και 104 αυτά για τις ε, πολύ πρόσφατα κατατεθεί στις τροπολογίες που ακόμα δεν έχουμε συζητήσει. Ευχαριστώ βεβαίω όλες και όλους τους κοιόδης συζητητές με τους οποίους συνεργάστηκα στενά και προφορικά αλλά και με ανταλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναμένω με ενδιαφέρον τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ κύριε Μάσιν. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν και ορισμένες τροπολογίες της Επιτροπής Αλίας που εγκρίνονται αυτόματα διότι εμπίπτουν στο άρθρο 50 της ε, ενισχυμένης συνεργασίας. Η Ζητώ συγγνώμη, ε, ε, είναι η πρώτη μου έκθεση και ίσως παρέψα να το πω. Σύμφωνα με το άρθρο 50, πράγματι η Επιτροπή Αλίας έχει κάνει συζητήσεις μαζί μου, αλλά και από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάρχει μια γνωμοδότηση δεν θα περιλάβω πολλά από αυτά, πολλές από τις διατυπώσεις τους, γιατί θα σήμαινε διπλασιασμό, πλεονασμό, επικάλυψη. Είναι πράγματα δηλαδή τα οποία λέμε ήδη εμείς. Και ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου και να υποστηρίξετε τις θέσεις μου. Εγώ το λέω αυτό. Γιατί τροπολογίες 7 ε, και 12 δεν θα τις ψηφίσουμε, γιατί ήδη συμφωνήσαμε. Τώρα για τις γνωμοδοτήσεις μπορούμε να ψηφίσουμε. Αυτά ως προς τη διαδικασία. Κύριε Κουμουτσάκο. Δύο γενικές σκέψεις στην αρχή. Ε, πιστεύω όπως και οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε ότι η ισχυρή θαλάσσια παράδοση είναι ένα μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη, ειδικά στις σημερινές πολύ αντίξωες οικονομικές συνθήκες. Είναι μονόδρομος λοιπόν κύριε Πρόεδρε να αναπτύξουμε όσο περισσότερο μπορούμε το μεγάλο δυναμικό των διάφορων τομέων θαλάσσας δραστηριότητα. Έτσι θα υπηρετήσουμε το συνολικό στρατηγικό μας στόχο για βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη, για απασχόληση και καινοτομία. Πιστεύω λοιπόν ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική υπηρετεί αυτούς τους στόχους. Προσφέρει ένα συνεκτικό πλαίσιο για διατομιακή δράση στις ευρωπαϊκές θάλασσες. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να στηριχθούν και να ενισχυθούν δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν κυρίως τη θαλάσσια διακυβέρνηση, τη θαλάσσια επιτήρηση αλλά και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα για την ουσία της έκθεσης που συζητάμε σήμερα. Άλλωστε θα έχουμε ευκαιρίες στο δρόμο προς την υιοθέτησή της από την Ολομέλεια να ξανασυζητήσουμε ε, επί της ουσίας. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω την κυρία Μάισνερ για την ειλικρινή και άοκνη συνεργασία μας. Ε, πιστεύω ότι επιτύχαμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συναδέλφους σκιώδεις ηγητές και των άλλων πολιτικών ομάδων. Συμφωνούμε με τις προτάσεις συμβιβασμού που έχουν κατατεθεί, αλλά πέραν αυτών ε, ελπίζω ότι θα έχετε ήδη δει ε, έναν αριθμό προφορικών τροπολογιών που έχω καταθέσει στην προσπάθειά μου να επιτευχθεί το ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός συνένεσης. Και ε, με την εισηγήτρια αλλά και μεταξύ των, των συναδέλφων. Οι προφορικές αυτές τροπολογίες αφορούν τις τροπολογίες 39, 51, 52, 55, 63, 83, 84, 97, 104 και το Recital E. Όλες αυτές οι προφορικές τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Να γίνει σεβαστή η επιθυμία της εισηγήτριας για μια όσο το δυνατόν συντομότερη, συνεκτικότερη και περιεκτικότερη έκθεση. Αφενός, λοιπόν, έπρεπε να, ε, να σεβαστώ αυτή την επιθυμία της συγκήτριας και δεύτερον, να λάβω υπόψη μου κρίσιμες και σημαντικές τροπολογίες που κατέθεσαν από συναδέλφους, ειδικά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, έχω καταθέσει και προτείνω τις, ε, τροπολογίες, ε, τις προφορικές αυτές τροπολογίες στις οποίες, ε, στις οποίες αναφέρθηκα μόλις πριν. Είναι όλες γραμμένες, όλη η προσπάθεια είναι να γίνουν συντομότερα ε, τα κείμενα, διατηρώντας τις ενδιαφέρουσες ιδέες που υπήρχαν σε αυτές. Ε, ενδεχομένως ε, μέχρι και την ε, αυριανή ψηφοφορία να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη ώστε το κείμενο να γίνει ακόμα πιο συντομότερο. Θα ήθελα όμως κλείνοντας κύριε Πρόεδρε να αναφερθώ με ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην τροπολογία 77 του συναδέλφου κυρίου Φλάνκενστάιν. Ε, η οποία αναφέρεται στο γνωστό σε όλους ε, ζήτημα του SO2 levels. Η τροπολογία είναι 77, επαναλαμβάνω. Ε, αντιλαμβάνομαι την φιλοσοφία της τροπολογίας που έχει κατατεθεί από τον κύριο Φλακενστάιν, όμως θα πρέπει να τονίσω ότι το ζήτημα αυτό παρουσιάζει την εξής διάσταση και είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί και να την προσέξουμε όλοι. Τα ειδικά αυτά καύσιμα, τα ε, χαμηλής περιεκτικότητος θείου, είναι δυσέβρετα. Η, ποιότητα η ποσότητα που υπάρχει στην αγορά δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Αυτό το γεγονός καθιστά το καύσιμο αυτό πάρα πολύ ακριβό. Εάν λοιπόν εφαρμοστεί στο σύνολο της Ευρώπης η υποχρέωση για τέτοιου είδους καύσιμα, να χρησιμοποιούνται τέτοια είδους καύσιμα, υπάρχει ορατός και μεγάλος κίνδυνος να έχουμε modal shift, μια αλλαγή λοιπόν στον τρόπο μεταφοράς και αυτό να γίνει εις βάρος της, ε, της, ε, της short shipping, short sea shipping, της αλίας μικρών αποστάσεων και προς όφελος του, της οδικής μεταφοράς. Αυτό είναι κάτι που αντιβαίνει στη βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές και θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you, ευχαριστώ. Ο κύριος Αλκαντράουε. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη για τον Κλουτ Φλάκενστάιν, που είναι σκιώδη ηγητή, αλλά δυστυχώ σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγητρία και του σκιώδη ηγητέ για την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική βελτιώθηκε την περασμένη εβδομάδα η μορφή της έκθεσης, η δομή της και συμφωνήσαμε και για κάποια σημεία, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Θέλουμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, μια και, στην έκθεση για τη θαλάσσια στρατηγική μέχρι το 2018 αναφέρονται τέτοια σημεία, δεν χρειάζεται να τα παραλαμβάνουμε σε αυτή την έκθεση. Όπω είπε και η συγγήτρια, θέλει να επικεντρωθεί σε θέματα διακυβέρνηση και διοικητικών δομών και όχι σε λεπτομέρειε ανακλάδο. Επίσης, θέλει όλα τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζονται με το σωστό τρόπο και με καλύτερο συντονισμό. Πιστεύω ότι μετά την ψηφοφορία την αυριανή θα διαμορφωθεί μια πολύ καλή έκθεση. Έχουμε παρόλα αυτά κάποια σχόλια. Καταρχήν για την τροπολογία 27. Ακούσαμε από την εισηγήτρια ότι είναι υπέρ. Μας χαροποιεί αυτή η δήλωση γιατί ήταν ε, η τροπολογία του Κνούτ Φλακενστάιν, 27. Καλή τροπολογία που προσπαθεί να βελτιώσει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Θάλασσας. Για την τροπολογία 77, από ό,τι ξέρω, η συγκέντρια είναι υπέρ και είναι όντως πολύ σημαντική τροπολογία, αναφέρεται στις οριακές τιμές ε, για το θείο, πολύ, στα κάψιμα, διοξίδιο του θείου. Περίπλοκο το θέμα, τεχνικό, με τεράστιες όμως συνέπειες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν συνθήκες ε, θεμητού ανταγωνισμού, χάρη σε αυτή την τροπολογία, ώστε να εξισωθούν οι τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ισχύουν πιο φιλόδοξες οριακέ τιμές σε ορισμένες χώρες και σε άλλες όχι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια εξομοίωση και θεμητός ανταγωνισμός. Από ό,τι ξέρω, η εισηγήτρια είναι κατά της τροπολογίας 78 που καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ταχθούν σε διεθνές επίπεδο για θέσπιση υποχρεωτικής χρήσης πλοηγού στα ιδιαίτερως επικίνδυνα διεθνή ύδατα όπως είναι στη Βαλτική, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι πετρελαϊκών καταστροφών από πλοία, λέει η τροπολογία 78. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι αδύνατο να επιβάλλουμε υποχρεωτική χρήση πλοηγού στα διεθνή ύδατα. Αλλά αν ε, η πλειοψηφία των μελών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού είναι υπέρ αυτής της θέσπης υποχρεωτικής χρήσης πλοηγού, είναι δυνατό ένα τέτοιο μέτρο. Και πιστεύουμε ότι βελτιώνει την ασφάλεια αυτών των ε, θαλάσσιων οδών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν που θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση για κατά πόσο είναι δυνατό να καταστήσουμε υποχρεωτική τη χρήση πλοηγού σε διεθνή ύδατα. Μπορεί να μας απαντήσει γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές ε, λύσεις, έχουμε πρόβλημα με την συμβαστική τροπολογία ε. Εμείς πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες που αντικαθιστά η συμβαστική είναι καλύτερες από την ίδια τη συμβαστική τροπολογία. Εμείς προτιμούμε τις ε, επιμέρους τροπολογίες όλες τις, το πρασίνων, της Άλντε, της Γκούε, του ΕΛΚ. Δεν είμαστε υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας που τις αντικαθιστά. Και τέλος, για τις προφορικές τροπολογίες, για την ε συμβαστική τροπολογία. Τώρα, για τις προφορικές τροπολογίες, λάβαμε μια δέσμη προφορικών τροπολογιών του ΕΛΚ. Ε, μάλλον δεν είναι δύσκολο, δεν είναι πρόβλημα περισσότερες από αυτές. Βέβαια, υπευλήθησαν καθυστερημένα και δεν μπορούμε λίγες ώρες πριν, έστω και μια νύχτα πριν την ψηφοφορία, να τις αναλύσουμε διεξοδικά. Θα ζητήσω το πάντως από τον σκιώδη μας γιατί Κνούτ Φλέκενστάιν να τις μελετήσει. Πάντως θα προτιμούσα τέτοιου είδους τροπολογίες να υποβάλλονται εμπρόθεσμα πιο έγκαιρα και όχι τελευταία στιγμή όπως έγινε. Κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω κάποιες παρατηρήσεις και για την έκθεση και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Έχω μία πορεία για τις τροπολογίες 25-27 για την παράταση της εντολής για την έμσα. Και κάποιες ανησυχίες. Έχουμε την έμσα, και στην συμβαστική τροπολογία δεν ξέρω που θα πρέπει να μπει. Συμβαστική τροπολογία Β, για παράδειγμα, και το θέμα που δημιουργήθηκε με την κατάσταση στον κόλπο του Μεξικού Ε, ή σε περίπτωση ατυχημάτων που εξοκύλουν ε, δεξαμενόπλη για παράδειγμα. Από ό,τι θυμάμαι, είχαμε μια προσωρινή εξεταστική επιτροπή στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Μετά ένα ατύχημα με δεξαμενόπλιο στις δυτικές ακτές Γαλλίας και Ισπανίας. Και το μάθημα που αντλήσαμε από αυτό το πάθημα είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πολιτική επέμβαση. Θα πρέπει οι ανεξάρτητες αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν τι σχετικέ αποφάσεις. Αυτό είναι λοιπόν το ένα θέμα. Υπάρχει το θέμα των δεξαμενοπλοίων με διπλή κήτη, διπλό κέλυφος. Ε, το θέμα είναι με τις ε, γεωτρήσεις ε, στο βυθό, σε μεγάλο βάθος. Μιλάμε για το ίδιο βάθος ε, στη Βόρεια Θάλασσα και στον κόλπο του Μεξικού. Αυτή είναι μια απορία που έχω, γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική για γεωτρήσεις πετρελαίου. Αλλά για τι βάθος μιλάμε, ισχύει το ίδιο βάθος. Πάντω, όντως η κατάσταση στον κόλπο του Μεξικού είναι τραγική. Και νομίζω ότι οι δικές μα προδιαγραφέ είναι πολύ καλές ε, και ισχύουν για την πετρελαιοβιομηχανία στις δικές μας ε, ακτές και είδωτα. Τώρα για τις συμβαστικές τροπολογίες. Η κατάσταση έχει περιπλακεί κάπως. Βλέπω και τις τροπολογίες, βλέπω και τις συμβαστικές τροπολογίες και δεν καταλαβαίνω πάντα τι εξυπηρετεί η συμβαστική τροπολογία. Αυτό τον προβληματισμό ήθελα να εκθέσω. Θυμάστε την ε, προσωρινή εξεταστική επιτροπή, ήταν πολύ χρήσιμη. Σε ό,τι αφορά το, την τροπολογία 85 για την εμπορία εκπομπών, γιατί είχαμε το θέμα της, ε, ε, του αποκλεισμού της αεροπορίας. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουμε κατά αντίστοιχο για τη θάλασσα. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 29, τις ε, μακροπεριφέρειες. Όταν μιλούμε για τον Ατλαντικό ωκεανό, τι ακριβώς ε, μακροπροσέγγιση εννοούμε. Γιατί τις ορισμένες περιπτώσεις έχει νόημα, σε άλλες όμως όχι. Επίσης, ό,τι αφορά τις επενδύσεις ε, στα ναυπηγεία και την ανανέωση του στόλου. Αυτή ήταν η αρχική τροπολογία. Εμείς ε, στις νότιες χώρες Μεσογείου έχουμε προβλήματα από ό,τι στο βορρά. Το θέμα είναι πώς θα ενθαρρύνουμε την άνθηση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Και γνωρίζουμε ότι δεν προβλέπονται ενισχύσεις για τα ναυπηγεία. Παρ' όλα αυτά, η ναυπηγική βιομηχανία είναι πολύ ελκυστική και θα πρέπει να οθούμε τους νέους να στρέφονται προς εκεί. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, εγώ ως Βρετανία θα ενδιαφερόμουν για το τι θα έκανε μια τέτοια Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή στις ακτές της ε, Μεγάλης Βρετανίας. Φυσικά και θέλουμε περισσότερο συντονισμό και συνεργασία. Τώρα, αν χρειαζόμαστε πραγματικά μια Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, τι να σας πω, ίσως είναι ευχολόγιο περισσότερο αυτός ο κατάλογος. Γιατί έχουμε χωρικά ύδατα, έχουμε περιφερειακά ε, διεθνή ύδατα, δεν ξέρω αν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Η κυρία Μάισνερ προσπάθησε να καταλήξει σε συνετές συμβαστικές τροπολογίες. Μερικές παρά είναι μακροσκελής πάντως. Και τέλος για τα ειδικά μία για τις ακτές και ολοκληρώνω σε λίγο κύριε Πρόεδρε. Τι προπολογισμό έχουν αυτά τα ταμεία για τις ακτές, ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτών των κονδυλίων. Ούτως ή άλλως ε, τα κράτη-μέλη έχουν οικονομικά προβλήματα. Ίσως λοιπόν τα πενιχρά κονδύλια που διαθέτουμε καλό θα ήταν να τα χρησιμοποιούμε πιο σύνετα. Η κυρία Μάισνερ προσπάθησε να συμμαζέψει κάπως το κείμενο. Αλλά εγώ θα προτιμούσα μία πλούστερη προσέγγιση, τουλάχιστον για ορισμένε συμβαστικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και την εισηγήτρια. Κύριο Στέιλορ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δύο πολύ σύντομε ερωτήσει πρώτα απ' όλα σε εσά. Ίσως μία για εσά και μία για κάποιον άλλον ίσω. Όσον αφορά τη διαδικασία στην Ολομέλεια. θα θεωρηθεί στρατηγικού ενδιαφέροντος αυτή είναι η έκθεση και αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Όσον αφορά τη συμβαστική πρόταση Α, μήπως κάποιο θα μπορούσε να μου εξηγήσει ποια είναι η γαλάζια στρατηγική για την ανάπτυξη. Γιατί ε, κανένα δεν το έχει αναφέρει μέχρι στιγμή και πρέπει να σα πω ότι πολύ προσεκτικά τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ίσως ε, η συγγήτρια ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να ε, σας καλύψει πάντως ε, οποιαδήποτε έκθεση από εμά, κατά τη γνώμη μου, είναι στρατηγική σημασία. θα, θα φροντίσουμε λοιπόν να προσεχθεί δεόντως. Και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Ίσως πάντως η Συγγήτρια ή η Επιτροπή θα μπορούσαν να απαντήσουν το δεύτερο ερώτημα, όπως είπα και στην αρχή, κύριε Τέιλορ. Κύριε Συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι, ναι. Αν είστε σύντομο, ναι. Ναι, μπορείτε να συνεχίσετε. Να ευχαριστήσω την κυρία Μάισνερ, λοιπόν. Και χαίρομαι που βλέπω ότι οι πράσινοι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν το ψήφισμα. Ε ε, ε, ε, όπως το βλέπουμε εμείς, παρόλο που καταλαβαίνω τις ανησυχίες για την καθυστερημένη υποβολή όλων των τροπολογιών, που πραγματικά δεν είχαμε το χρόνο να εξετάσουμε ε, δεόντως. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την 85 και για το γεγονό ότι θα υπάρξει χωριστή ψήφο. Γιατί εκεί μιλάμε για ολοκληρωμένου στόχου μείωση ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο ε, σε σχέση με το όραμα για, το 2000, για την Ευρώπη 2020. Και επίση έχουμε το δεύτερο σκέλο, και εδώ χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί η κυρία Μάισνερ ε, υποστηρίζει αυτό το σύστημα εμπορίας των εκπομπών ως ε, παράδειγμα ενός ε, εργαλείου οικονομικής προέλευσης για τη μείωση των εκπομπών. Ένα παράδειγμα, Πρόεδρε, είναι έτσι και βεβαίως δεν είναι το μοναδικό στοιχείο προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερο, στη συνάντηση με την εισηγήτρια και τους Κιώδης ακούσαμε τις ανησυχίες των συναδέλφων όσον αφορά ε, την αυθυλία σε επικίνδυνες περιοχές, με επικίνδυνα φορτία σε ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές και απαγόρευση για διέλευση, ενδεχόμενη απαγόρευση. Ελπίζουμε όμως ε, ότι, θα έχουμε μια, ότι η αναθεωρημένη διατύπωση που μιλά για αποφυγή προβλημάτων από τέτοια πλοία θα ε, ε θα τύχει της υποστήριξης. και τέλος, ε, συμφωνούμε με τη συμφωνία να, ε, να, να υιοθετήσουμε εν μέρη την 4α ε, και κυρίως εκεί όπου ε, ε αναφέρεται η, δυνατότητα επιλογής από το μορατόριουμ για αυτές τις, αυτές τις διαδικασίες άντλησης κτλ. Επίση και για τον καθαρισμό της θαλάσσης από τις τα κτλ. Ευχαριστούμε κύριο Γκρός. Αν θα μπορούσατε βεβαίω ε, να είστε στον ε, πιο σύντομο, θα είμαστε ευγνώμονε. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πληροφορία που έχω είναι ότι οι στόχοι που έχουμε καθορίσει για τον Βόρειο, για την Βόρεια Ευρώπη, του 0,1 δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν. Και ότι ενδέχεται να υπάρξει, με, να υπάρξει μετακίνηση φορτίων από τη θάλασσα στα φορτηγά. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα κάποια εξήγηση. Αυτά για την ώρα. Thank you, Σα Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Μάισνελ για την εργασία της και ε, για τις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες που όπως είπε ο κύριος Αλκαντράουι ε, αποτελούν βελτίωση του κειμένου. Θα ήθελα Χωρί να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία 29. Στην τροπολογία μου. Από ό,τι κατάλαβα, η εισηγήτρια έχει κάποιε επιφυλάξει όσον αφορά ε, κάποια συγκεκριμένα τμήματα τη τροπολογία. Και αναφέρομαι στις συνδυασμένες μεταφορές που αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να υποστηρίξουμε την ιδέα αυτή, διότι αυτό που θέλουμε είναι να αναπτύξουμε αυτούς τους μικρούς θαλάσσιους διαδρόμους. Αν όμως δεν εξασφαλίσουμε τις συνδυασμένες μεταφορές, τις διατροπικέ μεταφορέ, τότε ποτέ δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τι θαλάσσιε αυτέ μεταφορέ ε, στο βαθμό που θα έπρεπε. Γι' αυτό ζητώ από την εισηγήτρια να επαναξετάσει το ζήτημα αυτό. Και να υποστηρίξει αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριο ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πιο σύντομο από ό,τι σκόπευα, γιατί η κυρία Φώστερ με κάλυψε μεγάλο βαθμό. Αν επιτρέπετε, ορισμένες, ε, ορισμένα σχόλια ε, και σας λέω το εξή, έτσι κάπως σκόρπια. Εξετάζοντας τις τροπολογίες, φαίνεται ότι αυτό το οποίο λείπει είναι ορισμένα ζητήματα που θα έπρεπε να αποτελούν μέρος μιας θαλάσσιας πολιτικής. Μία τροπολογία ε, έτσι με, μεγάλο, με, με, μεγάλο, με πολύ γενικό τρόπο αναφέρει το θέμα τη πειρατείας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Όχι μόνο στο κέρα της Αφρικής, αλλά ε, και στι ακτέ τη Ευρώπη, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό με εκπλήσει ιδιαίτερα ε, που δεν αναφέρεται το ζήτημα αυτό. Ένα άλλο συναφέ ζήτημα έχει να κάνει με τη θαλάσσια ασφάλεια. Και αυτό δεν αναφέρεται. Ε, δεν αναφέρεται τίποτα ε, που να παραπέμπει σε μια πρωτοβουλία παρόμοια με την πρωτοβουλία για τι ασφαλεί λιμένε. Κάτι άλλο, το οποίο λάβει τη απουσία του, είναι ο ρόλο του Frontex, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περιοχή τη Μεσογείου διότι γνωρίζουμε ότι ε, ε, ε το Frontex ακριβώ αντιμετωπίζει το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και δεν βλέπω ε, κα, κανένα, καμία αναφορά στο σώμα αυτό. Και κάτι άλλο, Πρόεδρε, όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Πάρα πολλέ τροπολογίε αναφέρονται στην ανάγκη για χρηματοδότηση. Για σημαντικά θέματα όπω την αυπηγική βιομηχανία κτλ. Και πρέπει να σα πω ότι με δυσκολεύει ιδιαίτερα το θέμα αυτό, γιατί παραπέμπει σε, προστατευ... σε... σε καταστάσει προστατευτισμού. Όπω είπε η κυρία Φώστερ, η χρηματοδότηση που απαιτείται φαίνεται ότι είναι όλο και μεγαλύτερη. Όταν όμως ταυτόχρονα Όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάζονται να προβαίνουν σε περικοπέ του εθνικού του προπολογισμού. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι σαν να ζούμε στα σύννεφα. Ζητάμε όλο και περισσότερη χρηματοδότηση ε, ε για διάφορα τμήματα της, ε, ε, των θαλάσσιων μεταφορών και δεν καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα. Και κάτι άλλο. Ε, εδώ θέλω να πω το εξή. Κυρίω ορισμένε τροπολογίε από του πράσινου με παραξενεύουν. Εκεί όπου ζητούνται ε, εναλλακτικέ ε, μορφέ ενέργεια. Ε, ολική ενέργεια. τι να σα πω, με τα πανιά δεν, δεν χρησιμοποιούμε την ελληνική ενέργεια, έτσι κι αλλιώ. Οπότε τι να κάνουμε, να γυρίσουμε προς τα πίσω ε, στα, στις Τριήρες και σε άλλα πλοία ας πούμε. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιούν σκλάβους δηλαδή που θα κάνουν το κουπί. Μα εδώ θα ερχόμαστε θα έχουμε πρόβλημα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όταν είχαμε ε, αυτές, τις, αυτές τις λέμβους με τα κουπιά, οι δίκοι είχαν δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή. Να μην ξαναγυρίζουμε και προς τα πίσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη μου άφηξη, γιατί έτσι Ήμουν γενή προ την εισηγήτρια. Δεν μπόρεσα να ακούσω ούτε την εισηγήτρια, ούτε το σκιώδη εισηγητή τη ομάδα μα. Αλλά δυστυχώ δεν καταλαβαίνει από αυρότητα η πολιτική αεροπορία. Πάντω οι τροπολογίε που είχαμε καταθέσει νομίζω ότι έτυχαν θερμής υποστήριξης. Οπότε και οι ανησυχία μα καλύφθηκαν και διασκεδάστηκαν από την τελική μορφή τη έκθεση. Και αυτό χάρη στι προσπάθειε και τη εισηγήτρια και του σκιώδους συγκεκριτή της ομάδας μου. Βέβαια, υπάρχουν ακόμη κάποιες δυσκολίες, αλλά δεν έχω αρκετό χρόνο για να τις αναπτύξω. Ε, με το 77 έχουμε πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είναι διακριτική η μεταχείριση που προτείνεται. Γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η ρήπαση, τόσο αυστηρότερες πρέπει να είναι και οι προδιαγραφέ που απαιτούμε. Τώρα για το ταμείο για τις ακτές, να ιδρυθεί αλλά όχι βάρος των ε, υπαρχών των ταμείων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Από αυτή την άποψη οι τροπολογίες 30 και 35 και 34 είναι καλές, αλλά οι τροπολογίες 31, 32 και 33, παρόλο που είναι τις συγγήτριες, είναι κάπως ε, ασυνεπής κατά τη γνώμη μου σε σχέση με, τη, το γενικό ήρμο της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τεγκάντες Πασκουάλ. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δύο θέματα που έχω υποβάλει και ως τροπολογίες. 75 που αναφέρεται σε δύσκολες θαλάσσιες περιοχές και που ζητεί άλλη μια φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μια ξεκάθαρη ανάλυση. Δεν είμαστε μόνο Επιτροπή Μεταφορών, είμαστε και τουρισμού. Μπορεί κανείς να προβάλλει διάφορα οικολογικά επιχείρηματα, όταν όμως συμβαίνουν βαριά ναυτικά ατυχήματα που προκαλούν καταστροφές και προκαλούν βαρύτατες ζημίες και στον τουρισμό, διότι είναι βαρύτατη την ρήπανση των παραλιών, ε, πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Τώρα επίσης 77 και 78 μιλώ για IMO και MARPOL και στο παράρτημα 6 ιδιαίτερος όπου λέει ότι από το 2010 στα ευρωπαϊκά λιμάνια θα πρέπει να εκλείεται μόνο 0,1% θείων Αλλά όπως ε, ε, ο κ. Γκρός που τα είπε σωστά, χρειαζόμαστε και μια μελέτη επιπτώσεων του τι θα σημαίνει δηλαδή το 0,1%. Και ε, αλλού έχουμε κάνει τροπολογία και είπαμε ότι πρέπει να γίνουν προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εμπειρογνώμονες όλοι λένε 0,5% θείο περιεκτικό ταφείο δηλαδή στα καύσιμα, αλλά έχει καθοριστεί από το 2020. Άρα εδώ πρέπει να ισχύσουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και γι' αυτό ζητώ οι συνάδελφοι να επανεξετάσουν ολόκληρο αυτό το θέμα των τροπολογιών αυτών. Παρακαλώ κύριε Κουμουτσάκο, ζητήσατε πάλι το λόγο. Πολύ ευχαρίστως, άρα παρακαλώ σύντομος. Κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία 78 του κύριου Φράγκενστάιν όσον αφορά την υποχρεωτική ε, πλοήγηση ε, σε ιδιαίτερα επικίνδυνα η διεθνή ύδατα. Ε, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι δεν είναι ρεαλιστική αυτή η πρόταση. δεν, μπορεί, δεν, δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια πολιτική υποχρεωτικής πλοήγησης σε ποια ύδατα, πώς θα καθοριστούν, με ποια κριτήρια, αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, τι καθιστά επικίνδυνα κάποια ύδατα και ακίνδυνα κάποια άλλα. Ε, νομίζω ότι ε, ορθώς η ε, συγκήτρια εισηγείται αρνητικά στη συγκεκριμένη τροπολογία. Ευχαριστώ. Thank you. If I could just... Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα σύντομο σχόλιο. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Είναι σχετικά με την απόφαση τη Regional AMO για την περιεκτικότητα σε θείο διότι ανεξαρτήτως προθέσεων η πραγματικότητα είναι ότι προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ βορρά και νότου της Ένωσης. Για αυτό το λόγο πρέπει να εξεταστεί το θέμα. Το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα συζητήθηκε και στην Αμβέρσα σε επίπεδο υπουργών θα αναμένω από την Επιτροπή, λοιπόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μας πει με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πάντως, οι χώρες μέλη το υπέγραψαν. Οφείλω να το πω αυτό. Γιατί γνωρίζετε ότι ορισμένε φορέ κάνουν πράγματα που για μα είναι ανεξήγητα. Και, να, λοιπόν, ένα τέτοιο συνέβη και τώρα. Άρα, το φταίξιμο το έχουν οι χώρες μέλη. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά αυτά που προκαλούνται, προκαλούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναμένω λοιπόν από εισηγήτρια και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν κάποιες ιδέες. Βέβαια υπάρχει ανάγκη να διατηρηθούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού. ο κύριος Πένα νομίζω είναι από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, ω εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή σα για την πολύ θετική έκθεση, το σχέδιο έκθεση και απέναντι στι πρωτοβουλίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν θετική και συγχαρητήρια κυρία Μάισνερ για την πολύ αξιόλογη σας έκθεση. Θα ήθελα εν συντομία να σχολιάσω τα πιο σημαντικά θέματα στη συζήτηση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα με την ιδέα ότι θα πρέπει στις ε, μελλοντικές μας πρωτοβουλίες για την πολιτική της θάλασσας θα πρέπει να τις εντάξουμε στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της ανακοίνωσης για την ε, ε, Ευρώπη του 2020. Θα πρέπει να δώσουμε πολιτική προτεραιότητα στις διάφορες πρωτοβουλίες και θα είναι πολύ πιο εύκολο να δώσουμε τέτοια πολιτική προτεραιότητα εφόσον ενταχθούν στο γενικότερο πλαίσιο της Ευρώπης του 2020. Μερικές από τις προτάσεις σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό γιατί συμφωνείτε και με τη γενική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν υποβάλλετε και συγκεκριμένες προτάσεις, τις σημειώνουμε προσεκτικά και θα τις εξετάσουμε με τη δέουσα προσοχή για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτές. Για παράδειγμα το θαλάσσιο έρασμος, το να το αέρασμα στην αυτιλία. Θα το εξετάσουμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτή και βιώσιμη μια τέτοια πρόταση. Συμφωνούμε επίσης απόλυτα με την απήχηση που είχε στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη το δυστύχημα στο κόλπο του Μεξικού. Και μάλιστα οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή προβαίνουν σε μια εξονυχιστική ανάλυση τη ισχύουσα νομοθεσία για να διαπιστώσουν κατά πόσο ισχύουσα αυτή η νομοθεσία είναι σε θέση να καλύψει ταχύτατα και επαρκώς τέτοιου είδους καταστροφές. Και το ζήτημα της χρηματοδότησης της θαλάσσης πολιτικής είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα στις 29 του μηνός, μεθαύριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει ένα σχέδιο κανονισμού που θα θεσπίσει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο για την θαλάσσια πολιτική για την τριετία 2011, 2012 και 2013. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε αυτή την πρόταση ενδελεχέστερα στην Επιτροπή σας. Και χάρη στην πρόταση αυτή θα προβλεφθούν τα επαρκή δημοσιονομικά μέτρα για τη συνέχιση πολλών πρωτοβουλειών μας σε θέματα θαλάσσιας πολιτικής. Σημειώνουμε και την πρόταση για την σύσταση και ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής Υπηρεσίας είναι ένα είδος ε, παράτασης ε, της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Θάλασσας, κάτι που προϋποθέτει έλεγχο επιπτώσεων, μελέτη επιπτώσεων προηγούμενη. Πάντως ε, θα εξετάσουμε κατά πόσο είναι εφικτή μια τέτοια πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα οι Γενικές Διευθύνσεις ΜΑΡΕ, Περιβάλλοντος, και κλίματος προσπαθούν να συντονίσουν τις πολιτικές τους ώστε οι διάφορες πρωτοβουλίες για θέματα στρατηγικής της θάλασσας να λαμβάνουν υπόψη και τις προτεραιότητές μας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Φυσικά και θέλουμε μια φιλοπεριβαλλοντική ναυτιλία και σημειώνουμε τις σχετικές προτάσεις και ιδέες σας. Θα εξετάσουμε το κατά πόσο είναι εφικτές στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα, στο πρόγραμμα εργασίας μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει και μια στρατηγική για τον τουρισμό στις ακτές και μία από τις ερωτήσεις ε, που υποβάλλατε σε σχέση με την τροπολογία 78, το κατά πόσο είναι δυνατόν λοιπόν να επιβάλλουμε υποχρεωτικά την, την παρουσία σε επικίνδυνες ζώνες. Τη σημειώνουμε, θα την υποβάλουμε στην αρμόδια υπηρεσία και θα σας ε, δώσουμε διεξοδική απάντηση το αργότερο αύριο. Σήμερα το βράδυ θα την αναλύσουμε και αύριο το πρωί θα σας δώσουμε μια απάντηση. Τώρα γιατί δεν μιλούμε για πειρατεία στην ε, θαλάσσια πολιτική. Ένας από τους τρεις βασικούς άξονες της ε, πολιτικής των θαλασσών αφορά τον έλεγχο και την ολοκληρωμένη επιτήρηση της θάλασσες. Και στο πλαίσιο αυτό, το έργο της Frontex αποκτά κεφαλαιόδη σημασία. Και φυσικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αν αναφερθείτε και σε αυτή την πρωτοβουλία στην έκθεσή σας. Αυτά κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Mr. Mr. is ρωτήσω, η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ γνωρίζει τα προβλήματα με, το, ε, με, με, με, με το, την του του θείου στα βόρεια, στη Βόρεια Θάλασσα. Γιατί δεν αναφερθήκατε καθόλου στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, βεβαίω γνωρίζουμε πολύ το πρόβλημα αυτό και οι διάφορε ε, υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζουν θέση την οποία θα κοινοποιήσουμε στην Επιτροπή σε όσο τον πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ, η συγκίτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τα σχόλια των συναδέλφων μου. Θα αρχίσω από το τέλος. Επειδή το άφησα ε, έξω αυτό, διότι ήξερα ότι πολλοί θα αναφερθούν στο προβληματισμό αυτό περί θείου. Εγώ η ίδια κατοικώ στην βόρεια ακτή της Γερμανίας, η Βαλτική θάλασσα είναι κοντά στην περιοχή μου και γνωρίζω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια, στην οποία συμμετέχω κι εγώ, να βρεθεί λύση. Είναι καλό που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα ε, υποβάλει σχετική πρόταση. Μέχρι το 2015 δεν μπορώ, προλαβαίνουμε να τηρήσουμε τους στόχους αυτούς. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν αυτό, κανείς όμως δεν βγαίνει να το πει δημοσία. Γι' αυτό πάντως θεωρώ ότι είναι σωστό να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε κάποια λύση. Θα προσπαθήσω τώρα να απαντήσω στις διάφορες ε, τροπολογίες. Αλλά μην ανησυχείτε κύριε Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ σε όλες. Αυτά που είπε ο ο Φλέκενστάιν, τα είπα ήδη για την 75 και 77. Την νέα αυτή παραλλαγή μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Δεν θέλουμε, αλλά ούτε το λέμε και μέσα ότι μέχρι το 2015 θέλουμε να είναι το 1% ναι, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι τελώς παράλογο και δεν γίνεται. Να δούμε μόνο πώς μπορούμε να αποφύγουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, διότι βεβαίως ναυσιπλοεία δεν είναι μόνο στη Βαλτική θάλασσα, αλλά παντού. Και γι' αυτό θέλουμε η Βαλτική να γίνει ακόμα πιο ε, φιλική προς το περιβάλλον και όπως είπα σε όλες τις θάλασσες, από τη Βαλτική μέχρι τη Μεσόγειο και μέχρι τον Εύξηνο Πόντο. Το είπε και ο ε, Πρόεδρος distortion of competition είπε. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να αποφευθεί. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι και εμείς ως Επιτροπή του Κοινοβουλίου μπορούμε να δώσουμε κάποιο παράδειγμα με ε, την βοήθεια βέβαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για ορισμένα άλλα πράγματα τώρα. Σχετικά με την υποχρέωση για πλοηγούς. Μου είπε η Κομισιόν ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να επιληθεί φαίνεται πως είναι τροπολογία, όπως ε, μου είπε ο συνάδελφός μου, των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Δεν είμαι όμως εμπειρογνώμων για το θέμα. Θα δοθεί όμως απάντηση από την Κομισιόν. Πάλι αυτό μου είπαν. Εάν είναι δυνατόν πρέπει να το ξανασκεφτούμε, ναι. Εγώ πάντως τα ρωτήσει ειδικού, είχα μορφώσει την άποψη ότι δεν γίνεται. Τώρα η κυρία Φώστερ, αλλά η κυρία Φώστερ είναι απασχολημένη από ό,τι βλέπω. Κυρία Φώστερ της ομάδας ECR, είπατε ότι είναι κάπως φλίαρη η έκθεση. Ναι, εγώ παρόλα αυτά προσπάθησα να την κάνω σύντομη, αλλά συμβαίνει αυτό όταν υπάρχει πλήθος τροπολογιών που όλες έχουν την αξία τους, είναι δύσκολο μετά να τη συγχωνεύσει κανείς σε συμβιβασμούς. Και έτσι το κείμενο καμιά φορά γίνεται ιδιαίτερα μακροσκελέ. Μάλιστα, εγώ αναγκάζομαι να απορρίψω ορισμένε, γιατί μη θα γινόταν το κείμενο ακόμα μακροσκελέστερο αλλά επί της ουσίας προσπαθώ βέβαια να κρατήσω τα διάφορα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά ε, την ακτοφυλακή, τα είπε και η κυρία Φώστερ, ήδη προηγουμένως η Κομισιόν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είχε ε, συμφωνήσει η Κομισιόν να εξετάσει την συμπερίληψη της ακτοφυλακής, αλλά δεν έγινε τελικά αυτό. Ο κ. Πίτσικ, ο προκατοχό μου, το είχε αναφέρει. Blue Cross Strategy, ρωτήσατε τι είναι. Δεν θα τη βρείτε βέβαια ε, στο λεξικό, αλλά εγώ το έχω δει πολλές φορές αυτό, τον όρο. Και σημαίνει για μένα ανάπτυξη στον τομέα της θάλασσας. Υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό στις παράκτιες περιοχές και βεβαίως για την δημιουργία απασχόλησης. Αλλά βέβαια δεν είναι πραγματική ορολογία της αγγλικής γλώσσας αυτό, αλλά ας το υποστηρίξουμε. Είναι πάντως καλό σύνθημα εντό εισαγωγικών. Για το prohibitive shipping θα το κοιτάξω όπως είπατε, είναι κάτι διαφορετικό. Ε, θα δω τώρα μια στιγμή στις σημειώσεις μου αν λησμόνησα κάτι, γιατί βλέπω ότι ο πρόεδρος αρχίζει και ανυπομονεί. Αλλά πάντως νομίζω ότι είπα τα περισσότερα. Ευχαριστώ πάντως όλες και όλους για την εντατική συνεργασία. Α, ναι, και κάτι ακόμη για την Frontex. Είπατε ότι δεν περιλαμβάνεται. Περιλαμβάνεται. Frontex και πειρατεία, αλλά όχι τόσο εκτεταμένα. Γιατί σκέφτηκα ότι άλλα θέματα είναι πιο σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάλι λοιπόν όλες και όλους και χαίρομαι που σύντομα θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε το κείμενο ώστε μετά να μπορέσει να προχωρήσει και να εφαρμοστεί από την Κομισιόν. Τώρα έχω το εξή πρόβλημα. Ορισμένοι επιθυμούν να λάβουν και πάλι τον λόγο και όλοι μου λένε ότι θα είναι σύντομοι. Γκρός πρώτα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Βλέπω στην τροπολογία 77, εγώ τουλάχιστον την ερμηνεύω ως εξή που προτείνει ο κ. Φλέκενστάιν, ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία διάκριση μεταξύ Βορρά και Νότου και ότι ο Νότος θα πρέπει και αυτός να έχει και να χρησιμοποιεί ό,τι χρησιμοποιείται στον Βορρά. Εάν αυτός είναι ο στόχος, αλλά αν η εισηγήτρια κατανοεί κάτι διαφορετικό, τότε α το εξηγήσει, α το δηλώσει τώρα και α το εξηγήσει. Γιατί από αυτή την εξήγηση θα επηρεαστεί και η στάση που θα τηρήσουμε στην ψηφοφορία για την τροπολογία αυτή. Κύριε Σάλκαντράουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί τη διαδικασία, όσον αφορά την 78, την τροπολογία 78, για την υποχρεωτική παρουσία πιλότου στα ε, πλοηγού, στα επικίνδυνα ύδατα. Από ό,τι κατάλαβα, η εισηγήτρια θέλει την άποψη τη Επιτροπή. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή τη είπε ότι η απάντηση θα δοθεί αύριο το απόγευμα. Αλλά αυτό θα, γίνει, αυτό θα είναι μετά την ψηφοφορία. Πώ μπορούμε λοιπόν εμεί να αξιολογήσουμε το ζήτημα αυτό τώρα, ή λοιπόν να συμφωνήσουμε να επανέλθουμε ε, στην Ολομέλεια, όσον αφορά το σημείο αυτό, και να μπορέσουμε εκεί να ε, υποβάλουμε τροπολογία, αν είναι δυνατόν, αφού ακούσουμε δηλαδή την άποψη τη Επιτροπή. Ή δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Τροπολογία. Αύριο θα πάρουμε απόφαση την τροπολογία 78. Και αν στο μεταξύ έχουμε πληροφορίε μέχρι την Ολομέλεια, κάθε ομάδα ε, έχει το δικαίωμα να υποβάλει προφορική τροπολογία. Στην Ολομέλεια. Αυτό ήθελα να πω όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ο κύριο Γκρό. Νομίζω ότι εδώ ε, ίσως θα πρέπει ε, να έχουμε την ίδια αντίληψη, ε, ε, να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που κάνουμε και, στα, και στο νότιο τμήμα των θαλασσών και όχι το αντίστροφο. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά τα, τις, βόρειες, τις, βόρειες, τις βόρειες θάλασσες ε, έχουν προσυπογράψει τα κράτη-μέλη ε, και το ξέρει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα, αν έρθει σε επαφή με τον Επίτροπο, αλλά και με τους ε, Υπουργούς, ε, όλοι συμφωνούν στο ότι διεπράχθη ένα λάθος. Χρησιμοποιώ διπλωματική διατύπωση αυτή τη πάντως έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι προήλθε από, το, από τον IMO, από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, ότι είναι περιφερειακή η, η απόφαση. Και είναι ε, δεν είναι συνηθισμένο να παίρνει τόσο γρήγορα αποφάσει ο ΑΕΜΟ. Συνήθω χρειάζονται χρόνια και χρόνια. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν γίνονται βεβαιασμένα οι αποφάσει, ε, γίνονται λάθη. Θέλετε, κυρία Μάισνερ, να επανέλθετε. Ε, κυρία Μάισνερ, ναι, έχω κάνει μια σχετική έρευνα και γνωρίζω ότι όντω η Γερμανία έχει προχωρήσει διότι θεωρεί ότι είναι απαραίτητο αυτό επειδή η Βαλτική είναι τόσο επιβαρημένη. Αλλά οι ίδιοι οι Γερμανοί γνωρίζουν ότι δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένεται να μπορέσουν να τηρήσουν τους ε, στόχους αυτούς όλες οι χώρες. Γι' αυτό πρέπει να δούμε ότι ναι, όντως προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, αλλά βέβαια όχι αμέσως. Για τον κύριο Γκρός. Ο κύριος Φλέκενστάιν δεν είναι παρόν δυστυχώς, αλλά έχω συζητήσει μαζί του κατ' επανάληψη και σκεφτήκαμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα και γνωρίζω τι εννοεί. Ίσως είναι και θέμα μετάφρασης βέβαια, αλλά στο δεύτερο μέρος λέει ότι θα πρέπει να προστατεύονται όλες οι ακτές. Και, γι αυτό να μην, και για να μην υπάρξει distortion of competition, όπως είπε ο Πρόεδρος. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ό,τι ακριβώς ισχύει στη Βαλτική θάλασσα πρέπει να ισχύει και στη Μεσόγειο. Εγώ πάντως αυτά καταλαβαίνω ότι εννοεί ο κ. Φλέκενστάιν. Καλώς. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία την αυριανή ψηφοφορία που θα αρχίσει στις 9 και 10. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξη που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους. Ο κύριος Ρόιτ απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Είναι έξω από την αίθουσα, θα τον φέρουμε μέσα για να αρχίσει η ανταλλαγή απόψε. Okay, ladies and gentlemen, those who wish to hold their meetings. Παρακαλώ, όσοι έχουν συνομιλίες ιδιωτικές, να περάσουν εκτός αιθούσης. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον κύριο ρόιτε από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση που θα μας κάνει την εισαγωγή για την αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους. Μάλιστα έχει την καλοσύνη να μας φέρει και σχετικές διαφάνειες για να βλέπουμε και κάτι την ώρα που θα μιλάει. Κύριε Ρόιτα, έχετε το λόγο. Thanks a lot, uh, and, uh, Ευχαριστώ. Και καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι ιδιαίτερος που θα σας παρουσιάσω της προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους. Όπως ξέρετε, η πρόταση αυτή εγκρίθηκε πριν από 10 ημέρες. Και μάλιστα εσείς ήσασταν ε, στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και με την κριτική σας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Και τώρα μπορείτε να εξετάσετε πια την απόφαση, πολύ σημαντικό νομοθετικό πακέτο, που ευελπιστούμε ότι θα μας επιτρέψει να περάσουμε στην υλοποίηση του ονείρου μας για τον ενιαίο χώρο ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, που δεν θα είναι πια ένας ευσεβής πόθος και ένα όνειρο που θα φαίνεται στα χαρτιά, αλλά θα αποκτήσει σάρκα και οστά. Πριν από μία επταετία υιοθετήσαμε από κοινού την πρώτη μερική απελευθέρωση των σιδηροδρόμων και το άνοιγμά τους προς τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και μία τριετία μετά ολοκληρώσαμε τη διαδικασία αυτή, γιατί μας δέσμευαν πολλές προθεσμίες και όπως βλέπουμε από τα στατιστικά στοιχεία, και αυτό θα σας δείξω ορισμένες διαφάνειες, δεν φτάσαμε ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ε, όγκου μεριδίου στην αγορά και διείσδυσης ε, νέων ενδιαφερομένων. Οι διαφάνειες αυτές δείχνουν σε κάποιο βαθμό και την επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα των σιδηροδρόμων. Η πρώτη διαφάνεια δείχνει τις τάσεις σε ό,τι αφορά τις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων την περίοδο 2000-2007. Ορισμένες χώρες παρουσιάζουν άνθηση της μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει μια καθοδική πορεία. Οπότε δεν υπάρχει μια σταθερότητα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των μεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η Ιρλανδία Λουξεμβούργο, Γαλλία. Θα σας ε, δώσουμε πάντως τις ε, διαφάνειες. Δεύτερη διαφάνεια που περιλέγθηκε και στο ψηφισμά σας για την περίοδο 95-2007 το μερίδιο των σιδηροδρόμων στην μεταφορά εμπορευμάτων. Μέχρι το 2000 είχαμε μια πτωτική πορεία και τώρα πια έχω μια σταθεροποίηση του μεριδίου των σιδηροδρόμων, αλλά σταθεροποίηση σε πολύ χαμηλό επίπεδο δυστυχώς. Τρίτη διαφάνεια, τα μερίδια αγορών, αυτό που λέμε non-incumbent rail freight operators για τα τέλη του 2008. Και εδώ βλέπουμε τρεις κατηγορίες. Την κατηγορία του 40%, του 20% και μετά την τρίτη κατηγορία από μηδενικό ποσοστό μέχρι 20%. Και βλέπετε ότι η νομοθεσία μας, το νομοθετικό αυτό πακέτο έχει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα στα κράτη-μέλη. Σε γενικέ γραμμές λοιπόν, το άνοιγμα των αγορών ίσως βοήθησε για να αναστείλουμε την φωτική πορεία των σιδηροδρόμων, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αισθέθηκε με μεγάλη επιτυχία, όπως περιμέναμε πριν από μια δεκαετία κατά την εισαγωγή αυτού του πακέτου. Και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι ο ανταγωνισμός, το δεύτερο είναι η κανονιστική επίβλεψη και το τρίτο η χρηματοδότηση και η χρέωση των υποδομών. Για τον αθέμητο ανταγωνισμό τι έχετε να πείτε, τον εντάσσω στην πρώτη κατηγορία, στον πρώτο άξονα. Πρόσβαση στις αγορές. Είναι καθόδες αυτό το θέμα, βλέπετε τα στοιχεία για τους νέους α, παρόχους, αλλά και για τους α, ε, γνωστούς παρόχους. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Ισχύουν μεροληπτικοί κανόνες εις βάρος των νέων παρόχων. Επίσης έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις και παραδείγματα που μας δείχνουν πολύ δυσάρεστες πρακτικές ό,τι φορά την πρόσβαση στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και διακριτική μεταχείριση εις βάρος των νέων παρόχων. Επίσης, η διακριτική μεταχείριση μεταξύ incumbent και non-incumbent. Δεν υπάρχουν εναλλακτικέ ό,τι αφορά τους σταθμούς, ε, οι προβλήματα και στην πληροφορική αλλά και στο θέμα της ε, χρέωσης και της έκδοσης εισιτήριων. Για όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ανταγωνισμό. Δεύτερον, έχουμε τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά γιατί δεν λειτουργούν. Ανακύπτει το εύλογο ερώτημα. Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό, αλλά δεν υπάρχει αρκετή ανεξαρτησία. Δεν έχουν αρκετές αρμοδιότητες αυτές οι αρχές για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Πολύ συχνά οι θυμιστικές αυτές αρχές δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες, έχουν πολύ περιορισμένη εντολή, δεν μπορούν να κάνουν εκτεταμένες έρευνες, δεν μπορούν να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους με επιβολή κυρώσεων ή προστήμων. Πολύ συχνά το δικαστικό σύστημα είναι υπέρ των ιστορικών παρόχων και η βραδιπορία των των διαδικαστικών διαδικασιών είναι εις βάρος των νέων παρόχων, γιατί πολλές φορές ε, περνάει μια πενταετία, μια δεκαετία για την έκδοση μιας απόφασης. Πολύ συχνά η ρυθμιστική αρχή πάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών, άρα υπάρχει ένας έλεγχος των ιστορικών παρόχων, incumbent, και υπάρχει και θέμα σύγκρουσης συμφερόντων για συμβίβαστο. Και τέλος, πολύ σημαντικό επίσης θέμα, η ποιότητα των υποδομών. Δυστυχώς σε πολλές φορές μέλη οι υποδομές ε, παρακμάζουν, δεν υπάρχουν ποιοτικέ επενδύσεις, γιατί οι επενδύσεις στο σιδηροδρομικό κλάδο δεν είναι αρκετά, αρκετά εκκληστικές ούτε για τους ιστορικούς ε, παρόχους, ούτε για τους νέους, τους νέους ερχόμενους. Επίσης δεν υπάρχει σωστή δημοσιονομική, σωστός δημοσιονομικός σχεδιασμός για τις επενδύσεις στις ε, υποδομές και υπάρχουν και οι πρακτικές ότι αφορά τη χρέωση που είναι τόσο αποκλίνωσης και τόσο ασταθείς που δεν δίνουν κίνητρα στους επενδυτές για να επενδύσουν τις υποδομές. Ένα παράδειγμα για τη χρέωση. Και τι, μην με ρωτήσετε τι σημαίνει 960 cross φρέιτ. Οι διαφορές πάντως μεταξύ των κρατών μελών είναι τεράστιες. Και αυτές οι διαφορές επιδεινώνουν την κατάσταση. Ένα άλλο εύλογο ερώτημα που ανακύπτει. Εσείς το απαντήσετε, θα απαντήσω και εγώ από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παραβιάσεις ή αλλαγή, ε, μάλλον ε, διώξεις για τις παραβιάσεις ή αλλαγή της νομοθεσίας. Και τα δύο χρειάζονται. Το σιδηροδρομικό πακέτο υιοθετήθηκε το 2000 ε, και παρατάθηκε μέχρι το 2007. Ορισμένα προβλήματα οφειλόταν σε ατελή μεταφορά τη οδηγία στην Εθνική Νομοθεσία. Γι' αυτό και πριν τι θερινέ διακοπέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή κατά 13 κρατών μελών και εξετάζουμε και τις περιπτώσεις 9 ακόμη χωρών μελών για να δούμε μήπως θα πρέπει και εις βάρος αυτών να λάβουμε κάποια μέτρα και να κινητοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες. Πολλές φορές εξακολουθούν να προστατεύουν του, το κρατικό, τους κρατικούς παρόχους, ενώ η, η πλήρης εφαρμογή των οδηγιών του πρώτου πακέτου υποχρεώνει σε σημαντικό άνοιγμα των αγορών. Το τελευταίο πακέτο για τους σιδηροδρόμους συνοδεύτηκε από ένα ερμηνευτικό σημείωμα. Είχαμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη για την ερμηνεία συγκεκριμένων διατάξεων. Αυτά έγιναν το 2007 και το 2008 καταλήξαμε σε παραδοχή της διαφωνίας μας ό,τι φορά την ερμηνεία της ύπαρξης ε, νομοθεσίας. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό έδειξε και η εμπειρία μας τις τελευταίες δεκαετίες, γνωρίζουμε ότι κάποια τμήματα του νομοθετικού πακέτου θα πρέπει να εξυγχρονιστούν, να αποσαφινιστούν και να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά. Γι' αυτό και έχουμε μια παράλληλη διαδικασία. Εκτό από τι προσφυγέ της βάρος των κρατών μελών, προωθούμε και κάποιε νομοθετικέ αλλαγέ του πακέτου. Το πρώτο στοιχείο αυτής της ε, αλλαγής ή της αναδιατύπωσης αφορά την απλοποίηση της δέσμησης αυτών των νομοθετικών μέτρων. Αυτή τη στιγμή έχουμε 12 διαφορετικά νομικά κείμενα για τους σιδηροδρόμους. Και φυσικά και τις ε, συνθήκες διεύρυνσης προσπαθούμε να τα ενοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πακέτο για τους σιδηροδρόμους. Στόχος της αναδιατύπωσης αυτής είναι και η διευκρίνηση ορισμένων διατάξεων και η βελτιστοποίηση της εφαρμογής άλλων διατάξεων. Και θα επανέλθω εδώ στι ε, τρει διαφορετικέ κατηγορίε που σα ανέφερα και προηγουμένω. Καταρχήν, σε θέματα ανταγωνισμού. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια των συνθηκών πρόσβαση στην αγορά των σιδηροδρόμων. Με, με δηλώσεις ε, δικτύου που θα είναι πιο ενδελεχείς από τους διαχειριστές ε, των υποδομών. Θέλουμε να βελτιώσουμε την εγγυημένη πρόσβαση στις σιδηροδρομικές μεταφορές και για το εμπόριο επιβατών και για το εμπόριο εμπορευμάτων με συγκεκριμένους κανόνες για σύγκρουση συμφερόντων και αποφυγή διακριτικών πρακτικών. Σε ό,τι αφορά την ρυθμιστική επίβλεψη, επισκόπηση, προτείνουμε παράταση των αρμοδιοτήτων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και για τις συναφείς με τους σιδηροδρόμους υπηρεσίες, ε, ενίσχυση της ανεξαρτησίας αυτών των ρυθμιστικών αρχών από τα άλλα κρατικά σώματα και φορείς και ταυτόχρονα τον εφοδιασμό τους ε, με καλύτερα μέσα για την επιβολή των νομοθετικών μέτρων. Κυρώσεις, ε, πρόστιμα και δυνατότητα έρευνας των παραβιάσεων. Και επίσης θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα κανονιστική και μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αριθμιστικών αρχών, προκειμένου να μην καταλήξουμε με τεράστιες διαφορές ό,τι αφορά τα θέματα χρέωσης, πρόσβασης στις, υποδομ... στις υποδομές κτλ. Και τέλος, αλλά πολύ σημαντικό θέμα, θέλουμε να προωθήσουμε το θέμα του δημοσιονομικού σχεδιασμού και για τις υποδομές. Θέλουμε να υποχρεώσουμε κατά κάποιο τρόπο τα κράτη-μέλη να χαράξουν μακροπρόθεσμες εθνικές στρατηγικές, πολιετής ε, ε, συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών και των διαχειριστών των υποδομών, χρηματοδότηση και επιβράβευση της απόδοσης, και στα θέματα της χρέωσης ασχοληθήκαμε με το θέμα της, του εσωτερικού υπολογισμού του εξωτερικού κόστους, ε, αντιμετώπιση του, της συγχωρήπανσης και ένα σύστημα για να δώσουμε στους παρόχους που χρησιμοποιούν μηχανισμού ε, μηχανισμούς ERTMS να λαμβάνουν κάποιες εκπτώσεις ότι αφορά τη χρήση του δικτύου. Αυτά είναι δύο στοιχεία για την εσωτερική, εσωτερικό υπολογισμό του εξωτερικού κόστους. Επίσης, ε, προτείνουμε μία ε, συνολική αξιολόγηση αντικτύπου, που βεβαίως την έχετε και οι συναδελφοί μου Βασκαβέλ Καστελέτη και λοιπά βρίσκονται εδώ σήμερα ε, και, και άλλοι συνάδελφοι βρίσκονται εδώ, αλλά και στο μέλλον θα μπορέσουν να σας εξηγήσουν όλα τα διάφορα στοιχεία αυτή τη αξιολόγηση αντικτύπου. Είμαστε πεπισμένοι ότι το διοικητικό άχθος από τα νέα μέτρα είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ωφέλη της δέσμευση. Και νομίζω ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να το υποστηρίξουμε και απαντώντα σε λεπτομερή στοιχεία. Δύο παρατηρήσει θα ήθελα να κάνω. Μάλλον τρει. Για να τελειώσω ε, την πρώτη μου εισαγωγική παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα, το άνοιγμα των χωρίων επιβατικών αγορών δεν το συμπεριλάβαμε στην πρόταση αναδιατύπωσης. Είναι πολύπλοκο ζήτημα. που σαφώς συνεπάγεται την, την αξιολόγηση ιδιαίτερα πολύπλοκων ζητημάτων, όπως για παράδειγμα σύνδεση με τον κανονισμό OSP, ε, τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά ο αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής, ο κύριος Κάλλας, μας ε, ε, ε απευθύνει έκκληση και είναι σαφές ότι μέχρι τέλος του 2012 θα έχουμε φτάσει τα διάφορα ζητήματα. Άρα και ενδεχομένως και τον ε, κανονισμό για τις δημόσιες υπηρεσίες θα έχουμε μια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί μόνο αν δεν ανοίξουμε την αγορά αυτή των επιβατικών μεταφορών, δεν θα έχουμε ε, ε, αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα του ενιαίου στερεοδομικού χώρου. Και όσον αφορά ε, την ολοκληρωμένη διαχείριση, εδώ θα γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο των μεταφορών, αλλά και τις ενέργειες και τα Και θυμάμαι ε, τον διαχωρισμό, ε, το unbundling και στον τομέα της ενέργειας ε, τι έγινε. Καλύτερα λοιπόν και εδώ να εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα ζητήματα και να ε, είμαστε σίγουροι ότι και το δικαστήριο θα ακολουθήσει την ερμηνεία που, θα, δίνουμε εμεί. Ε, να, δούμε, ε, να, λάβ, να λύσουμε τα διδάγματα από το διαχωρισμό στον τομέα της ενέργειας, να δούμε ε, το θέμα της αμεροληψίας του ε, ε, διαχειριστή, να δούμε όμως και σε σχέση με τις διαδικασίες επί παραβάση που έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή. Να μην δώσουμε την εντύπωση ότι υποχωρούμε. Αν τα πράγματα είναι καλά, να έχουμε το θάρρος και να πούμε πριν από 10 χρόνια δεν τα αντιμετωπίσαμε σε... όπως θα έπρεπε, ας το κάνουμε τώρα. Βεβαίω, αυτή η στρατηγική ασχολείται με ορισμένα τμήματα ε, του ενιαίου συνδρομικού χώρου. Πρέπει να εξετάσουμε και άλλα ζητήματα όπως το θέμα της ε, διαλειτουργικότητας, ε, ε, το θέμα του οργανισμού των σιδηροδρόμων, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα εξετάζουμε με ιδιαίτερα εντατικό τρόπο και θα υποβάλουμε ξεχωριστές προτάσεις. Μάλλον μέσα στον επόμενο χρόνο. Συνολικά πάντως πιστεύω ότι όταν θα έχουν ε, προχωρήσει και οι συζητήσει πάνω στι συγκεκριμένε προτάσει και με εσά και με το Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη, πιστεύω πάντω ότι τελικά αυτή η δέσμη θα αποτελέσει ένα ουσιώδε στοιχείο ε, του οράματο οράματος του Αντιπρόεδρου Κάλλας για τον ενιαίο ε, ε, χώρο στους ιδεοδρόμους, ε, ε, ένα όραμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι έχετε και στο σκηνοβούλιο. Αυτά είναι οι δυσαγωγείς και είμαι έτοιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις. ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Ρόιτερ. Όπως καταλαβαίνετε, έχω πολλούς ομιλητές στο κατάλογό μου. Να υπενθυμίσω όμως τα μέλη ότι Αν σας καλύψει κάποιος συνάδελφός δεν χρειάζεται να επαναλάβετε και εσείς την ερώτηση. Ε, το θέμα είναι να λεφθούν τα πάντα, όχι και από όλους. Ε, έχουμε μια ώρα περίπου για συζήτηση. Ε, πριν τους νοηστές, ξεκινώ με το ΕΛ και τον κύριο Γκρός. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, παρουσίαση αυτή. Είναι ιδιαίτερα θετική, είναι ε, ε, ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της αναδιατύπωσης αυτής. Έχουμε όμω κάποιε ανησυχίε. Αλλά είναι αλήθεια ότι συνολικά βλέπουμε το ζήτημα θετικά. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Θα έλεγα, κάπω ηρωνικά μου επιτρέπετε, ότι εδώ ε, δοκιμάζουμε ένα νέο φάρμακο, ε, ένα φάρμακο ε, το οποίο ε, στην ουσία το έφτιαξε ο ασθενής. Εδώ βρισκόμαστε δηλαδή απέναντι σε κάτι το οποίο είναι κάπως περίεργο και παράδοξο. Έχουμε δηλαδή μία σειρά από κυρώσεις και μία σειρά από τροπολογίες που υποβάλλουμε εδώ. και σε τελευταία ανάλυση, αν δεν εφαρμόσουμε όλα αυτά, τι νόημα θα έχουν. Δηλαδή, ε, εδώ, κοιτώντα το, το, το, το, σύστημα του ευρώμου στην Ευρώπη και τι αδυναμίε του συστήματο, αντιλαμβανόμαστε στην ουσία ότι πρόκειται για ένα τομέα ο οποίο, ένα κλάδο που αυτό που, που προσπαθεί να αποφύγει πάση θυσία είναι ο ανταγωνισμό με, με του υπόλοιπου τρόπου μεταφορά. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε και το θέμα και τι εποπτείε, το θέμα του ελέγχου εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να επανέλθουμε εδώ. Πρέπει οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο να έχει όσο περισσότερη πρόσβαση γίνεται σε ε, πηγές πληροφόρησης για να μπορούμε να θέτουμε ερωτήσεις ε, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία. Ε, γιατί δεν θα πρέπει δηλαδή να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου μετά από 5-6 χρόνια να δούμε ότι όλα αυτά είτε εφαρμόστηκαν λανθασμένα είτε δεν εφαρμόστηκαν καθόλου. Δεύτερον, διαλειτουργικότητα. Κοιτάξτε, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε ε, σε επίπεδο κανόνων και νομοθεσίας, αλλά εάν δεν δούμε το ζήτημα αυτό της διαλειτουργικότητας, παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες μας, τελικά δεν θα κάνουμε τίποτα. Γιατί όλα αυτά πρέπει, ε, οι νομοθετικέ πρωτοβουλίε θα πρέπει να ακολουθούνται και από την κατάλληλη ε, τεχνολογία. Δεν θα έχουμε διαφορετικά ένα ενιαίο χώρο στον τομέα των συνδρόμων. Αν εξακολουθήσουμε δηλαδή να έχουμε αυτά τα διαφορετικά συστήματα. Τέλο. Χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι ε, ουσιώδη σε τελευταία ανάλυση. Ε, όταν λοιπόν ε, κάνουμε την ανάλυση όλων αυτών και αναλύσουμε τα αρνητικά στοιχεία τα οποία μας δώσατε ε, και που ήδη είδαμε άλλωστε, αντιλαμβανόμαστε ότι ε, υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στις επιδόσεις και στο ποιος είναι φθηνός και στο ποιο είναι ακριβώς. Άρα η αλήθεια βρίσκεται κάπου αλλού. Και αυτό πρέπει να προκύψει από κάποια ανάλυση. Όταν μιλούμε για χρηματοδότηση, και γενικά για το κόστος στη μεταφορά εμπορευμάτων, είναι σημαντικό να γίνεται και σύγκριση και με μεταφορά προσώπων. Και βεβαίως να εξετάζεται τι επιθυμούν οι χώρες να επενδύσουν για τα επόμενα χρόνια. Επανέρχομαι στο θέμα των χρηματοδοτήσεων στις μεταφορές. Εδώ έχω να πω το εξής. Διαπίστωσα με ενδιαφέρον ότι στις μεταφορές και στον σιδηρόδρομο γίνονται ορισμένες επενδύσεις και από το Περιφερειακό Ταμείο, όχι μόνο από τα δικά μας, από τους δικούς μας πόρους εδώ της Επιτροπής Μεταφορών. Είναι σημαντικό λοιπόν οι χώρες να διαθέτουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρήματα, εφόσον βεβαίως εφαρμόζουν και τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διότι είναι παράλογο εμείς εδώ να νομοθετούμε και οι χώρες να χρησιμοποιούν τους ευρωπαϊκούς πόρους για να κάνουν πράγματα τα οποία στην ουσία αντιβαίνουν στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου. Άρα δηλαδή αποφεύγουν τελικά την διαλειτουργικότητα και αυτό μάλιστα με ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτό λοιπόν είναι μια σημαντική διάσταση του θέματος και ειδικά τώρα που μιλούμε για επαναδιατύπωση, αυτό το recast, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και ίσως μετά την εξέταση του θέματος να μπορέσουμε να εργαστούμε και με πιο, ε, συνεκτικό και πιο συνεπή τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκρός. Τώρα δώσουμε λόγο στον κύριο Άνικα Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, με, κοιτάξτε και εμείς πιστεύουμε ε, ιδιαίτερα ότι ε, οι, οι εμπορευματικές μεταφορές ε, με, με τους δρόμους ε, πρέπει να γίνουν με αυτόν τον τρόπο που αναφέρετε και εσείς με δυναμισμό, αναφέρετε τις δυσκολίες ε, αναφέρεται τα προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο συμμόρφωση. Άρα, σε τελευταία ανάλυση δεν υπάρχει θεμητό ανταγωνισμό στον ε, τομέα, πράγμα το οποίο ανακόπτει ε, την μελλοντική εξέλιξη αυτών των σιδηροδρομικών ζωνών στην Ευρώπη. Υπάρχουν προβλήματα ερμηνεία, άνισα μέτρα κτλ. Όλα αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε και θα πρέπει να δούμε μήπω θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε ορισμένε επιμέρου τροπολογίε και αλλαγέ σε ορισμένου τομεί. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, η νομοθεσία να είναι σαφέστατη και να επιτρέπει συγκεκριμένε συμφωνίε όσον αφορά το ποιο προτείνει ποιε υπηρεσίε, είτε σε επίπεδο, ε, σε επίπεδο μεταφορέων. Ε, παράδειγμα, η σταθμή ε, αποθήκευσης τι είναι, ε, ε, ε, ποιο έχει την ευθύνη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όσον αφορά για παράδειγμα αυτά τα παραδείγματα πρέπει να σκεφτούμε συνολικά το θέμα τη διαχείριση των δικτύων. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν πρέπει να εξεταστούν με λεπτομερή τρόπο και όσον αφορά την κανονιστική αρχή και εδώ οδεύεται προς την, την σωστή κατεύθυνση γιατί ε, μιλάτε για ενισχυμένε αρμοδιότητε, Αυτό που θα μα ενδιαφέρει τώρα εμάς να δούμε είναι ε, ε, λίγο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό και πιστεύουμε ότι εδώ μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, ιδιαίτερα για να καταλήξουμε σε ε, ανάλογε υποδομέ ε, με, με ανάλογε επιδόσει. Εσεί μιλάτε βεβαίω για μεγάλε διαφορέ όσον αφορά ε, τα τέλη πρόσβαση στα δίκτυα. Ε, ε, εδώ πρέπει λοιπόν να δούμε τη χρέωση κτλ. Εδώ πρέπει να δούμε ότι ε, η πτυχή αγορά δεν αρκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να ε, είμαστε ε, συνολικά ε, συνεπείς για να μπορέσουμε να, να εξασφαλίσουμε το μέλλον της πολιτικής αυτής. Κυρίως αναφορά τα προβλήματα αυτά τα οποία αναφέρει ο κύριος Κρός και που μάλλον θα ήθελα να φέρουν και άλλοι συνάδελφοι. Μιλώ για τη χρηματοδότηση και για τα ε, ε, νέα μέσα τα οποία θα επιτρέψουν τις επενδύσεις. Όταν μιλάμε για χρηματοδότηση, εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, εξασφαλίσουμε ανάλογες, ε, ε, ανάλογες συνθήκες ανάλογα με, τον τρόπο μεταφοράς, ευρωβινιέτα κτλ. Γιατί ε, θα πρέπει να έχουμε συνολική αντιμετώπιση για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Διαφορετικά δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Άλλο στοιχείο έχει να κάνει με την τεχνική διαλειτουργικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ο Ευρωπαϊκό Φορέα πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε και αυτό το οποίο θα ήθελα ε, ιδιαίτερα να ακούσω διαστόματό σα ε, είναι κατά πόσον και εσεί συμφωνείτε με το στόχο αυτό και κατά πόσο το χρονοδιάγραμμά σα έχετε προβλέψει κάτι παρόμοιο κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίση θα ήθελα μια συγκεκριμένη ιδέα για όλα τα μέτρα τα οποία ήδη έχουν ληφθεί ε, δια τη επιτροπολογία ή δια άλλη οδού για να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα και επίση θα ήθελα να μάθω τι προβλέπετε για τα επόμενα χρόνια προ την κατεύθυνση αυτή αυτά τα τρία στοιχεία θα πρέπει να εκθεστούν ω σύνολο. Λειτουργία τη αγορά, χρηματοδότητα, διαλειτουργικότητα σε τεχνικό επίπεδο. Κατά την άποψή μου, θα ήταν σφάλμα να ε, περιοριστούμε στην πρώτη πτυχή, δηλαδή στη λειτουργία τη αγορά. Κατά την άποψή μου, πρέπει να δούμε ταυτόχρονα και τι άλλε δύο διαστάσει του ε, ζητήματο αυτού. Τέλο, όσον αφορά ε, την ε, ενημέρωση εν ώψη τη μελλοντική απελευθέρωση των επιβατικών μεταφορών, εδώ πρέπει να σα πω ότι Υποστηρίζω την προσέγγιση σα. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τα αναλύσουμε όλα αυτά με πολύ μεγάλη προσοχή και άλλωστε αυτό συζητήθηκε και στα πλαίσια ε, τη ε, συμφωνία για την τρίτη δράση μισθονομικών μέτρων. Είχαμε πει ότι πρώτα ε, απαιτείται ε, λεπτομερέστατη αξιολόγηση αντικτύπου και στα πλαίσια τη συζήτηση αυτή αυτό το είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε το κατά πόσον όλα αυτά θα γίνουν προ το όφελο και το συμφέρον του επιβάτη. Γιατί αυτό που θα πρέπει να αποτελεί γνώμονά μα όταν ε, ε ξεκινάμε τέτοιε περιπέτειες. Και πράγματι πρέπει να ξεκινάμε με αυτό το στόχο. Και να σας θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, μας ε, μιλήσατε για αυτή τη μελέτη. Ω ήδη να είναι αποτέλεσμα μια συμφωνία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε και στο στόχο. Ποιο είναι ο στόχο τη μελέτη αυτή, Γιατί αυτό είναι ουσιώδε και για τη συνέχιση της συζήτησης. Και κάποια στιγμή θα ήθελα μια, ε, ένα ενδελεχή κατάλογο των στοιχείων προτίθεστε να μελετήσετε έτσι ώστε να υπάρξει συνολική δυνατότητα αξιολόγηση. Ευχαριστούμε κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ. Είπατε να μην επαναλάβουμε τα όσα ήδη ελέγχθησαν. Θα προσπαθήσω λοιπόν. Πάντω κάτι που δεν ελέγχθη και που με απασχολεί ως νέο μέλος είναι ότι ναι μεν εγκρίθηκε το πακέτο, αλλά 21 χώρες μόνο έχουν, έχουν ε, εγκρίνει και δύο από αυτές δεν έχουν κάνει σιδηροδρόμους. Και αυτό που λέει ο κ. Γκρός σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις, σωστό είναι. Είναι σωστό αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έστειλε δηλαδή προειδοποιήσεις, ότι δηλαδή έχει εγκριθεί το πακέτο και πρέπει να εφαρμόζεται. Βεβαίω και χρειαζόμαστε απελευθέρωση των σιδηροδρόμων και ό,τι αφορά τα, τους ε, πόρους, αυτά που ήδη εγκρίναμε στην Σαραγώσα. Δεν έχουμε βέβαια χρήματα επαρκεί για, όλους τους, ε, για επενδύσεις σε όλους τους λεγόμενους διαδρόμους. Γι' αυτό χρηματοδοτούμε ιδίω διαμεθοριακά έργα. Και η διαλειτουργικότητα που δεν υπάρχει, διότι τα συστήματα δεν είναι συμβατά. Και εκεί δεν κινούνται οι χώρες μέλη. Εμείς πάντως ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε σε αυτά ακριβώς να, κάνουμε, να συμβάλλουμε. Αφενός πάντως πρέπει να λεχθεί ότι καμία χώρα, σχεδόν μόνο τέσσερις, δεν έπραξε ό,τι έπρεπε, αλλά και να κάνουμε και προτάσεις οι οποίες δεν θα αντιμετωπίσουν μόνο την αντίσταση των χωρών μελών, αλλά θα επιτρέψουν γενικά στο σιδηρόδρομο να προχωρήσει. Και όπως είπε και ο Επίτροπος, να πετύχουμε αυτό τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Έτσι είπε ο Επίτροπος και ελπίζω να μπορέσουμε να κινηθούμε προς τα εκεί να δούμε ποια βήματα είναι απαραίτητο να γίνουν. Συμφωνώ με τον κύριο Ελχαντράουι που λέει ότι θα ήθελε να μάθει ποιο νόημα έχει η μελέτη, δηλαδή τι υποτίθεται ότι θα εξετάσει η μελέτη που προτίθεται να αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ των Πρασίνων. Πέντε λεπτά, Μιχέλ. Γιατί. Μου το λες μόνο εμένα και, όχι στους άλλους. Καλά λοιπόν. Για τις ερμηνείες της, για την ερμηνεία μάλλον, ερμηνεία που δίνεται μάλλον στην διαφορετική ε, νομοθεσία. Εμείς θέλουμε διαχωρισμό του δικτύου από τη λειτουργία του. Και αυτό με τη σωστή ερμηνεία. Τώρα αυτό γίνεται, ποια είναι η άποψή σας. Γιατί περιμένουμε την απόφαση του δικαστήριου και δεν μπορούμε να πούμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί δεν λέμε και στη Γερμανία συγκεκριμένα ότι αυτό που κάνει αντίκειται στο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Διαφάνεια. Στο Βερολίνο πληρώνουν οι σιδηρόδρομοι τα διπλάσια από ό,τι στο Αμβούργο. Και το Αμβούργο τα διπλάσια από αυτά που ε, πληρώνονται ε, στον χώρο του Ρήνου και του Μάιν. Πρόσβαση. Και εδώ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, τα είπαμε και τελευταία. Η Γαλλία, για παράδειγμα, κατήργησε τον ε, φόρο επιχειρήσεων για τις δικές της επιχειρήσεις, για τις επιχειρήσεις τώρα των άλλων χωρών που κινούνται μέσα στην επικράτειά της παίρνει αυτό τον rolling stock tax. Μια στιγμή. Ναι. Αλλά είναι αδικία όμως διότι πληρώνουν και τον ΦΠΑ και τους υπόλοιπους φόρους και τα τέλη αυτά, την εισφορά αυτή δηλαδή που επιβάλλει η Γαλλία. Έχουμε έναν οργανισμό, ευρωπαϊκό οργανισμό, αλλά εφόσον υπάρχει αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός και οι εθνικοί οργανισμοί σιδηροδρόμων δεν συνεργάζονται, τότε δεν χρειάζεται ο ευρωπαϊκός. Ό,τι θα ρυθμίζει όμως ο ευρωπαϊκός οργανισμός δεν χρειάζεται να ρυθμίζουν οι εθνικοί. Αλλά εκεί έγκυται και μεγάλη αντίφαση. Τώρα, κρατικά κονδύλια για τις υποδομές Αυτά γίνονται, αυτά δίνονται μόνο υπέρ των δημοσίων οργανισμών, όχι για όλους. Και αυτό είναι, και αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ούτως ή άλλως υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός με άλλους φορείς ε, μεταφορών, ορισμένοι πλέον φόρο προστέμενης αξίας, άλλοι όχι και ούτω καθεξής. Και αυτό πρέπει να σας απασχολήσει. Με τη μεταφορά προσώπων στο σιδηρόδρομο στο τρίτο πακέτο των σιδηροδρόμων υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία και μόνο επειδή έγινε πέμπτη απόγευμα δεν είχαμε την απαραίτητη δική πλειοψηφία. Θα έχετε λοιπόν την υποστήριξη του Κοινοβουλίου γι' αυτό. Για το ΙΑΤΜΕΣ δεν είπατε τίποτα. Εδώ, εδώ εννοώ. Η Γερμανία απορρίπτει 23 εκατομμύρια. Να λάβει δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ΕΑΤΕΜΕΣ. Μα έχουν υπογράψει συμβάσεις. Οι άλλες χώρες γύρω-γύρω επενδύουν στο ΕΤΕΜΕΣ και η Γερμανία όχι. Ίσως, ίσως αυτό είναι μια προσπάθεια να απομακρύνει άλλους ανταγωνιστές. Για τα θέματα των επενδύσεων θεωρώ δεν είναι μόνο θέμα των, των χρημάτων και για τα τέσσερα μεγάλα έργα Μπρένερ, Λεόν, Τουρίνο και Μεσίνα κτλ εάν είναι σε 30 χρόνια έτοιμα κατά 40-50% εμένα δεν με ενδιαφέρει κανένα δεν πρόκειται να μας ωφελήσει. Στο Βερολίνο για παράδειγμα επενδύθηκαν δισεκατομμύρια για ένα νέο σύστημα ε, σιδηροδρομικών γραμμών και εν τέλει όλοι περνάνε μέχρι και 60% περισσότερο χρόνο στους ε, σιδηροδρόμους διότι ήταν εσφαλμένες οι επενδύσεις αυτές. Δεν αρκεί δηλαδή το μέγεθος των επενδύσεων για να δικαιολογήσει την επένδυση. Επίσης, στο πακέτο των σιδηροδρόμων είπαμε τότε ότι 40% το λιγότερο πρέπει να πάνε στον σιδηρόδρομο. Και είχε δώσει και θετική γνώμη τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Μπαρό τότε είχε ταχθεί υπέρ. Αλλά το Συμβούλιο δεν ασχολείται. Όμως εκεί βρίσκεται ομοχλός. Όσο δίνεται 60% στον δρόμο, στην, ε, στον αυτοκινητόδρομο και 40% στον σιδηρόδρομο, να μην σας εκπλήσει ότι δεν προχωρούμε. Αυτό είναι ο πραγματικός μοχλός. Και μπορούμε να πούμε και στις χώρες μέλη ότι αν θέλετε ευρωπαϊκά χρήματα, ναι, σας δίνουμε, αλλά για να κινηθείτε στη σωστή κατεύθυνση, όχι στη λάθος κατεύθυνση, γιατί τότε δεν σας υποστηρίξουμε. Αυτό θα είχε νόημα. Ο, ο, ο κανόνας 1370 αρχικά στην πρόταση περιλαμβάνονταν και οι σύνδρομικέ επιχειρήσει. και μετά εξαιρέθηκαν. Γιατί? α μην παραπονούνται τώρα, μην παραπονείστε μάλλον εσεί τώρα γιατί εσεί φταίτε στην Κομισιόν. Εμείς θέλαμε να σα υποστηρίξουμε. Τελικά όμω προέκυψε ένα παράξενο συμβιβασμό, εκεί χάθηκε μια ευκαιρία. Την πρόταση γκρό την υποστηρίζω και η νομοθετική έκθεση, κυρία Μάισνερ, πρέπει να προχωρήσει. Μιλεί μακριά από το μικρόφωνο κύριος Κράμερ, δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε καλά. Υπερβάλλω λέει, αλλά νομίζω ότι η πρόταση είναι ορθή και πολύ σύντομα θα το αντιληφθούν. Όσο όμως νομίζουν ότι θα μπορέσουν να λάβουν τα χρήματα και τους κάνουν θα τους κάνουν οι ίδιοι, θα συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο. Και τελευταίο, για να τηρήσω τα πέντε λεπτά μου, θα ωφελήσει αυτούς που κινούνται με το σιδηρόδρομο. Αυτό είναι και το κρίσιμο ερώτημα. Εάν εξετάζουμε μοναχά την αποδοτικότητα, την οικονομική αποδοτικότητα, θα χάνουμε στο σιδηρόδρομο. Εάν μειωθούν οι επιβάτες του σιδηρόδρομου κατά 25%, θα είναι καλύτερη σολισμή των τρένων. Εν πάση περιπτώσει, κινητικότητα είναι θεμελιώδες δικαίωμα και πρέπει να ενταχθεί στην κοινωνία. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι το μοναδικό κριτήριο αυτό η αποδοτικότητα. Εάν ορισμένε ιδεοδομικέ επιχειρήσει λένε ότι θα βάλουμε εμεί ένα ποσοστό για την επένδυση και τα υπόλοιπα θα τα βάλει το κράτο, δεν πάει καλά. Θα είχε νόημα εάν συν πλήν φτάνουν στο 0 ή έστω και μείον 5 ή μείον 6%. Χρειάζεται να, γίνει, να, χρειάζεται να προσεχθεί αυτό. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ η οικολογική διάσταση και η οικονομική βέβαια, αλλά μην λησμονούμε την κοινωνική διάσταση. Thank you. That's the Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το γύρο των συντονιστών, αλλά και πέντε ευρωβουλευτές ζήτησαν τον λόγο. Ο κύριος Βαντάλεν προσθέθηκε από τους συντηρητικούς στο γύρο των συντονιστών. Ευχαριστώ. Κύριε Ρόιτε, νομίζω ότι ήσταν πολύ μετριόφρον στα συμπεράσματά σας και πολύ μετριοπαθείς Είπατε ότι ίσως θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το άνοιγμα των σιδηροδρομικών αγορών διέκοψε την παρακμή των σιδηροδρόμων, αλλά δεν οδήγησε σε σημαντικότερη άνθηση. Ε, δεν είναι και ε, αρνητικό αυτό. Είναι αρκετά εντυπωσιακό. Θα μπορούσατε να είστε υπερήφανος, γιατί και το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών αυξήθηκε σε πολλές χώρες μέλη. Προτάθηκε τώρα μια διπλή προσέγγιση της αναδιατύπωσης και των διαδικασιών επί παραβάση κατά των κρατών μελών. Πώς όμως θα εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων του πρώτου νομοθετικού πακέτου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είστε πιο αυστηροί απέναντι στα κράτη-μέλη και να μην διστάσετε να ασκήσετε διαδικασίες επί παραβάση. Γιατί ήταν διαφορετική η μεταχείρισή σα απέναντι σε διάφορε χώρε. Δεν θα πρέπει να είστε πιο διστακτικοί απέναντι σε ορισμένες και πιο επίκης απέναντι σε άλλε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είστε εξίσου αυστηροί και απαιτητικοί από όλε και να τη σύρετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση που παραβιάζουν το πακέτο των νομοθετικών μέτρων. Κυρία Μάισνερ, είπατε ότι είναι πολύ θετικές οι εξελίξεις και εκφράσετε την επιθυμία σας να βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά είστε κυβερνών κόμμα. Θα πρέπει λοιπόν να πιάσετε τον τάβρα από τα κέρατα και να είστε πιο απαιτητικοί στην εφαρμογή. Στις κάτω χώρες, για παράδειγμα, ε, επιταχύναμε τη διαδικασία της απελευθέρωσης και διαπιστώνουμε ότι πολλοί πάροχοι που προσφέρουν υπηρεσίες με ανταγωνιστικές τιμές και με πολύ ε, καλύτερη ποιότητα είχαν επιτυχία. Γιατί λοιπόν δεν ε, προσπαθείτε να μας μιμηθείτε και στη Γερμανία. Ο κύριος Σρίκε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι και λακωνικός και να μην επαναλάβω τα όσα ακούσαμε μέχρι στιγμής. Μία γενική ε, παρατήρηση που απορρέει από την μικρή πύρα που έχω ως Ευρωβουλευτής. Όντως είναι αρκετά χρονοβόρες οι διαδικασίες, αλλά διαπιστώνω ότι το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο δεν απολυλειτούργησε. Οπότε θα υιοθετήσουμε τις παλιές μεθόδους, οπότε θα αντιμετωπίσουμε παρόμοια προβλήματα ή θα περάσουμε σε μια ανώτερη ταχύτητα και θα αναθεωρήσουμε τον τρόπο της μέχρι τώρα δράσης μας. Για παράδειγμα, το να επέβουμε στις επενδύσεις μέσω της χρηματοδότησης θα μας, επιτρέπει, θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δράσεων, αλλά γι' αυτό χρειάζεται πολύ πιο σημαντική επέμβαση στα διάφορα, παρέμβαση στα διάφορα ε, προγράμματα. 10 με 20%. Θα πρέπει επίσης να γίνει μια ιεράρχηση των διαφόρων σχεδίων και να φτάσουμε σε ποσοστά αποφασιστικής σημασίας, να βελτιώσουμε και τη χρηματοδότηση με τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανισμούς. Ίσως ε, να συστήσουμε και ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο. Βέβαια, αυτή η πρόταση ίσως θα προκαλέσει διαμαρτυρίες, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό που θα επιτρέπει την παρέμβαση όπου χρειάζεται. Αλλά υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί. Για παράδειγμα, εξωτερήκευση και αναζήτηση άλλων μηχανισμών επέμβαση. Πάντως, μας ενδιαφέρει ε, πιο δραστική επέμβαση στις υποδομές. Σε ό,τι αφορά την, αιρεσιμότητα. Ναι, να ενισχύσουμε τα προγράμματα με σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αλλά όχι ανεφόρων, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και επίση η επέμβαση υποδομέ θα επιτρέψει καλύτερη ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού χώρου. Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έλεγχο, ήταν ανεπαρκή μέχρι στιγμή. Και είναι πραγματικά ε, εντυπωσιακό ότι θα ασκήσετε διαδικασία επί παραβάση κατά 21, 21 ε, χωρών. Θα πρέπει λοιπόν ε, και τα νομοθετικά μέσα και τα υλικά μέσα να τα ενισχύσουμε. Και υπάρχει και το θέμα της ε, ευρωπαϊκής ρυθμίσης. Χρειαζόμαστε, εκτός από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, και ένα, μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Για τη διαλειτουργικότητα έχει τεράστια σημασία, γιατί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την υπεκφυγή των εθνικών ε, παρόχων για να αποφύγουμε τη δράση. Γιατί χρησιμοποιείται αυτό πολλές φορές ως άλοθη. Ο νομοθετικός έλεγχος θα πρέπει να εξυπηρετεί άμεσα τη διαλειτουργικότητα αν δεν βελτιώσουμε τη διαλειτουργικότητα, γιατί μιλήσαμε για τον οργανισμό, αλλά θα πρέπει ο οργανισμός να είναι και αυτός λειτουργικός. Επίσης, θα πρέπει να ξαναβάλουμε τους σιδηροδρόμους ε, στο γενικότερο θέμα των συνδυασμένων μεταφορών. Και τέλος, αυτή, αυτός ο κατατεμαχισμός σε διάφορα πακέτα και ο διαχωρισμός μεταξύ μεταφοράς επιβατών και μεταφοράς εμπορευμάτων μας οδηγεί σε μια απώλεια αποτελεσματικότητα, αλλά και σε μια αποδυνάμωση του πολιτικού μηνύματος που δίνουμε και σε έναν πολλαπλασιασμό των νομοθετικών ή κανονιστικών κολλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Και αντί να εχουμε δύο, τρία, τέσσερα πακετα καλύτερα να έχουμε ένα καλό πακέτο βιώσιμο και αυθεντικό. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω πράγματι να είμαι πάρα πολύ σύντομη για να επιτρέψω τους άλλους συναδέλφους να τοποθετηθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, διότι πράγματι ε, αυτή η δέσμη ε, και η αναδιατύπωσή της είναι ε, πάρα πολύ σημαντική για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συνομικού Δικτύου. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω και εγώ την ανάγκη ε, να ασχοληθούμε με τρεις δράσεις πάρα πολύ σημαντικές, δράσεις στις οποίες αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι. Να έχουμε αυτό το ολοκληρωμένο ε, συνδρομικό δίκτυο ε, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες Σημαίνει σίγουρα ενίσχυση ε, του ρόλου των εθνικών ευρωπαϊκών αρχών, το έχουμε ήδη πει στο παρελθόν, σίγουρα σημαίνει να ε, δημιουργήσουμε ε, και, τον, και την ενιαία κανονιστική αρχή, αλλά κυρίως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ε, διαχωρίσουμε τους μεταφορείς και αυτούς που διαχειρίζονται τις υπηρεσίε, τις υπόλοιπε. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι και δεν ξέρω πώς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την ανακλειστή του δικτύου, γιατί αυτό θα αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και που ε, ξεπερνάει την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σίγουρα δεν προ την ορθή κατεύθυνση. Βεβαίω, ε, θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα μέτρα. Ορισμένα ε, τα έχουμε ήδη αναφέρει, όπω για παράδειγμα η διαφάνεια των τελών για όλου του Ευρωπαίου πολίτε, η ενίσχυση τη διαλειτουργικότητα σε τεχνικό επίπεδο και βεβαίω το σημαντικό θέμα, το οποίο ήδη αποτελεί αντικείμενο εξέταση, το θέμα τη χρηματοδότηση των μεγάλων υποδομών μόνο με αυτόν τον τρόπο πάντως θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ε, ένα ε, χώρο των σιδεροδρόμων που να, είναι, αποτελεί μια εναλλακτική λύση ε, αλλά εξίσου σημαντική εναλλακτική λύση έναν των οδικών μεταφορών. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζασάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση καλωσορίζω τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνάδουμε την βελτίωση των σιδηροδρομικών ε, μεταφορών και υιοθετεί διατάξεις για να δημιουργήσουμε ένα, πραγματικό δημοσιονομικό σχεδιασμό χωρίς να υπερβαίνουμε ε, υπερβολικά στη ρύθμιση της αγοράς. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι παρόλο που δεν είναι πολύ σημαντικέ οι νομοθετικέ ρυθμίσει, προκύπτει από το έγγραφο ότι τα αποτελέσματα τη αναθεώρηση για τα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντικά και επιτείνουν τη γραφειοκρατία και τον έλεγχο στι σιδηροδρομικέ μεταφορέ. Για παράδειγμα, προβλέπονται συγκεκριμένε διατάξει στα παραρτήματα τη οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αρμόδια ε, για τις κατα κατά εκχώρηση πράξει και άρα προβλέπει, προ... καταλήγει σε αυθαίρετες διατάξεις. Νομίζω ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει πραγματικές προτάσεις για τη βελτίωση των μεταφορών. Γιατί δεν θα πρέπει να έχουμε διαφορετικά ποσοστά σε ό,τι αφορά την πρόσβαση. Ούτε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το retrofitting χρηματοδότηση. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε δυσαναλογία μεταξύ των πιο ισχυρών και των λιγότερο ισχυρών παρόχων. Η υπερβολική παρέμβαση στον τομέα εξαιτία της αναθεώρησης ε, προκύπτει από τα παραρτήματα της οδηγίας. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο άχθος για τις νομοθέτες και μπορούν ε, τα μέτρα αυτά, τα υπερβολικά αυτά μέτρα να μπλοκάρουν την αγορά. Αναφέρθηκε στι κατά παραχώρηση δράσει δράσεις και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά και το κόστος τη υπερβολική ρύθμιση ε, θα είναι τεράστιο για το σιδηροδρομικό κλάδο. Κάτι που θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρόμου σε σχέση με, άλλες, με άλλους τρόπους μεταφοράς. Um, Σας ευχαριστώ. Ε, και εγώ, κύριε Ρόιτερ, για την ε, παρουσίασή σας και θα ήθελα να σας ε, υποβάλω μια σειρά από ερωτήσεις. Προφανώς, οι επενδύσεις στις υγειονομικές επιδομές είναι ουσιώδους σημασίας για για να έχουμε πραγματικά ποιοτικέ υπηρεσίες στον τομέα των συνδρόμων. Και είναι ουσιώδους σημασία, αν θέλουμε να πείσουμε του επιβάτε αλλά και τι επιχειρήσει να ε, επιλέγουν τι ειρηνικέ μεταφορέ εναντί άλλων τρόπων μεταφορά. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται ποτέ ένα επιβάτη να επιλέξει το σιδηρόδρομο εάν, ε, του, ε, εάν κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα, θα χρειαστεί διπλάσιο χρόνο για να φτάσει στον προορισμό του. Γι' αυτό η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξή. Πώ. Ε, πώς θα, πώς, θα, πώς θα πείσετε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στις ε, μεταφορές, να προβούν σε εξυγχρόνιση των δικτύων τους και πώς θα αναπτυχθούν ε, νέες δομές που να επιτρέπουν την κυκλοφορία τρένων υψηλής ταχύτητας. Η ε, ο σιδηρόδρομος πάντα ε, ήταν παράγοντας προόδου. Ακριβώς γι' αυτό και πιστεύω το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και, πρέπει να πιστούν τα κράτη-μέλη να προβούν σε επενδύσεις. Κάτι άλλο τώρα. Ε, είπατε για το ERTMS και το γεγονός ότι ε, ε μπορεί και αναφερθήκατε στο θέμα της έκπτωσης. Να σας υπενθυμίσω το εξής. Πέρυσι, ε, στην τελευταία δημοπράτηση, ορισμένα σχέδια έγιναν δεκτά και άλλα όχι. Άρα, Ορισμένα σχέδια έγιναν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, άρα ορισμένοι ε, μεταφορείς, ε, ορισμένοι επιχειρηματίες βρίσκονται πιο μπροστά και άλλοι, ενώ άλλα σχέδια απορρίφθηκαν. Με αποτέλεσμα, οι τελευταίοι επιχειρηματίε να μην έχουν δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτίθεται να εξασφαλίσει την ισότιμη ε, συμμετοχή στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Τώρα, επιτρέψτε μου να πάρω και εγώ το λόγο και να κάνω ορισμένε παρατηρήσει, κύριε Ρότε, πριν απαντήσετε σε αυτά τα οποία ακούσατε, στι ερωτήσει που ακούσατε. Α, όχι, πρώτα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντεγκράντε Πασκάλ. Πασκουάλ, ευχαριστώ πρώτα, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Σα ευχαριστώ, κύριε Ρότε, για την παρουσία σα και θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτά που είπε ο συντονιστή μα, ο κύριο Γκρό. Η χρηματοδότηση πρέπει να έχει άμεση σχέση με το στόχο. Άρα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν οι επενδύσεις. Δεύτερον, ε, είναι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Άρα εδώ ε, δεν θα πρέπει μόνο τα ευρωπαϊκά όργανα να φέρουν την ευθύνη. Πρέπει να, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι, ε, ότι μερικές φορές ε, τα κράτη δεν μπορούν να, ε, να εκπληρώσουν τις, τους στόχους τους γιατί ακριβώς αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, όνειρο θερινής νύχτας είναι το, το όνειρο του κυρίου Κάλλας. πραγματικά, πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τη χώρα μου, για παράδειγμα, ε, εμεί θα είμαστε μια χώρα που έχει το μεγαλύτερο δίκτυο τρένων υψηλή ε, ε ταχύτητα ε, ε, στον κόσμο. Και όμω ταυτόχρονα οι εμπορευματικέ μεταφορέ βρίσκονται σε, πολύ χαμηλό επίπεδο. Απελευθέρωση λιμένων το ίδιο. Ε, πολυτροπικότητα τίποτα. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση πρέπει να δούμε όλο αυτό το θέμα με σαφή πολιτική βούληση. Τέλος, να πω το εξής. Μερικές φορές ε, οι, οι δυσκολίε δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πολιτική βούληση των κρατών. Γιατί, Γιατί είναι τα διασυνοριακά ζητήματα ε, τα οποία αφορούν ε, κοινέ ε, ε, αρμοδιότητε. Και εδώ θα πρέπει να υπακρυπνά η Επιτροπή για Συμμόρφωση. Τέλο, να σα πω το εξή όσον αφορά ε, τα διαδικαστικά θέματα ε, αναδιατύπωσης. Θεωρητικά ε, τροποποιείται μόνο αυτό το οποίο βρίσκεται σε παχιά γράμματα, αλλά σε τελευταία ανάλυση στην πράξη γίνονται άλλα ζητήματα γιατί ακριβώς πρέπει να υπάρχει συνέπεια και στο κείμενο. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι μόνο τροποποιούμε αυτό το οποίο αναφέρεται σαφώς αλλά μερικέ φορέ, εάν δεν, κάνουμε, αν δεν αλλάξουμε και το υπόλοιπο κείμενο, υπάρχουν ασάφειε και συνέπειε. Θέλω να πω, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Thank you, Mr. De Grandes. Uh, as I... Ευχαριστώ, κύριε Δεγκράντε Πασκουάλ. Κύριε Ρόιτερ, αυτό το όλο θέμα της πρώτης αναδιατύπωσης Ναι. Είναι σαν ένα παιχνίδι με τρένο. Και υπάρχει ατμομηχανία, αλλά τα βαγόνια πίσω δεν ακολουθούν πάντα. Και αυτό το πρόβλημα παρατηρούμε με πολλά κρατημέλη που πολλέ φορέ κολλησιεργούν και δεν ακολουθούν την ατμομηχανία που φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ε, δούμε λοιπόν τον τρόπο που αναπτύχθηκαν οι σιδηροδρομικές μεταφορέ, αυτό διαπιστώνουμε. Είπε ο κ. Δεγκράντες Πασκουάλ ότι η Ισπανία είναι η χώρα που έχει τα περισσότερα δίκτυα και τα περισσότερα χιλιόμετρα ε, τρένων υψηλής ταχύτητας. Βέβαια, οι περισσότεροι επιβάτες που χρησιμοποιούν τους σιδηροδρόμους δεν χρησιμοποιούν ε, τα τρένα υψηλής ταχύτητας, αλλά τους, ε, τα συμβατικά τρένα, που πολλές φορές είναι ε, χαρακτηρίζονται από φοβερή πολυκοσμία και είναι αυτά τα τρένα που παίρνει ο κόσμο για να πάει στη δουλειά του. Αυτέ τι μεταφορέ, αυτού του είδου τι σιδηροδρομικέ μεταφορέ θα πρέπει να βελτιώσουμε. Επίση, το θέμα τη ανεξαρτησία του διαχειριστή των υποδομών είναι ζωτική σημασία. Ορισμένα κράτη-μέλη ακόμη δεν έχουν ε, ε εφαρμόσει τον κανονισμό 91-440 που προβλέπει το διαχωρισμό των υποδομών από τον διαχειριστή του δικτύου. Και δυστυχώς ε, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι να υλοποιήσουμε αυτό το διαχωρισμό. Είμαι υπέρ της αύξησης των αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών, είμαι υπέρ της ε, αποτελεσματικότερης ε, εργασίας των ρυθμιστικών αρχών, αλλά θέλω οι ρυθμιστικές αρχές πραγματικά να ρυθμίζουν τα πράγματα και να μην διαχειρίζονται τι σιδηροδρομικέ μεταφορέ και τα σιδηροδρομικά δίκτυα. Και η πατρίδα μου είναι ένα παράδειγμα. Εκεί κατηγορούμε τη ρυθμιστική αρχή ότι προσπαθεί να διαχειριστεί του σιδηροδρόμους αντί να αφήσει του διαχειριστέ ε, να διαχειριστούν του σιδηροδρόμους και η ρυθμιστική αρχή να περιοριστεί στην αρμοδιότητα τη ρύθμισης. Δεν θα πρέπει να υπάρξει σύγχυση τέτοιων αρμοδιοτήτων. Σε ό,τι αφορά τη χρέωση τη πρόσβαση. είναι υπερβολικά αυτά τα τέλη πρόσβαση. Και ιδιαίτερα ισχύει αυτό για, το εμπόριο των, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Είναι σαν τη σταχτοπούτα η μεταφορά εμπορευμάτων και όχι σαν την ύφη ή το προνομιακό σκέλος. Στην Ευρώπη δίνουμε προτεραιότητα στην ε, μεταφορά επιβατών. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να αναχαιτήσουμε την ε, μεταφορά των εμπορευμάτων. Και αυτά τα παράπονα ακούω περισσότερα. Αν μια τρίτη χάσει το σλότ ε, μια μεταφορά εμπορευμάτων για παράδειγμα, αυτή ήταν μια κατηγορία κατά της Γαλλίας. Κατηγορία αβάσιμη, δεν, υπάρχει, δεν είναι τεκμηρωμένη. Αν λοιπόν χάσει το σλότ της τρίτης, παίρνει σλότ την Τετάρτη. Όχι αργότερα την ίδια μέρα, αλλά μία μέρα μετά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η κατηγορία κατά της Γαλλίας. Αν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει μια τέτοια πρακτική να σταματήσει. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι από τους προβληματικούς σειρμούς του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρόμου, αλλά είναι πραγματικά γελίο. Αν κανείς μεταφέρει εμπορεύματα από το Λονδίνο στο Καλέ, που είναι μια σύντομη απόσταση, μικρή απόσταση, θα πρέπει να περάσει από τρία διαφορετικά καθεστώτα χρέωση υποδομών για να πραγματοποιήσει αυτή τη μεταφορά. Έχουμε το Βρετανικό σύστημα στο κανάλι της Μάχης και από εκεί και πέρα το Γαλλικό σύστημα, αλλά και το ειδικό σύστημα του καναλιού της Μάχης, όσο περνάει κάτω από το κανάλι. Και υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας. Και αν χρειαστούν κάποιες αλλαγές, θα πρέπει να προηγηθεί διακυβερνητική συνδιάσκεψη. Για μία μικρή απόσταση παρόλα αυτά. Γιατί να μην μπορούμε να μεταφέρουμε εύκολα εμπορεύματα με τη σύραγγα της μάχης. Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένουμε προτάσεις για να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα αυτό. Και αυτό είναι το όνειρό μου, όπως έλεγε και ο Μάρτιν Λουθερ έχω ένα όνειρο και το... η δική μου για τις επαγγελίες είναι ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που μπορεί, θα μπορεί κανείς να περνάει τα σύνορα χωρίς ε, να το σταματάνε κάθε τρεις και λίγο. Ο Μάρτι Λούθερ Κίνγκ είπε ότι εκείνο είδε τη γη τη επαγγελία. Εγώ δυστυχώ δεν είμαι βέβαιος ότι την έχω αντικρίσει. Ευελπιστώ όμω ότι θα τη δω πριν πεθάνω. Αλλά βλέποντα ότι έχουν ήδη ασπρίσει τα μαλλιά μου, βλέπω ότι ο χρόνο περνάει και ίσω να μην προλάβω να τη δω. Αυτό θέλουμε λοιπόν, να προχωρήσουν οι σιδηρόδρομοι και να προχωρήσουν απρόσκοπτα. Γιατί πολύ συχνά εκπρόσωποι των σιδηροδρόμων έρχονται και τα συζητάμε και όλοι λένε ότι το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς, Όλοι είμαστε υπέρ τη. Εμεί είμαστε υπέρ τη απελευθέρωση, αλλά δεν είμαστε εμεί το πρόσκομα. Κάποιο όμω δημιουργεί πρόβλημα. Κάποιο θα πρέπει να είναι ο υπέτειο που αναχαιτίζει την πρόοδο. Και, και εγώ προέρχομαι από του σιδηροδρόμου και αγαπώ τις, ε, του σιδηροδρόμους και αν εγώ εκνευρίζομαι, φαντάζομαι πόσο εκνευρισμένοι θα είναι ε, άνθρωποι που δεν έχουν σχέση πραγματικά με τους σιδηροδρόμους, που δεν τους αγαπούν τόσο όσο εγώ. Πω πω, μετά από αυτή την γεμάτη πάθος έκκληση, τι να πω εγώ. Ας αρχίσω τέλος πάντων λέγοντας ότι ήδη από το 98, 99 και τέλη το 99 είχαμε την κοινή θέση για, το, για την πρώτη δέσμη των σιδηροδρόμων. Ε, μεγάλο τότε υπουργό προεδρεύοντα, τον κ. Γκίσο, και με την Επίτροπο τότε Λοϊόλα Παλάσιο καταφέραμε να φτιάξουμε τον πρώτο συμβιβασμό, μετά έφυγα από τις μεταφορές, επανήλθα και αν με επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, έχουν αλλάξει οι σιδηρόδρομοι τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν μέσα σε μια αγορά επιθυμούν να ανταγωνίζονται, άρα τότε φταίνει οι κυβερνήσεις, λέει ο Μπράιν. Λέμε καμιά φορά το αστείο ότι λειτουργούν οι σιδηροδρόμοι, αλλά το μόνο πρόβλημα που έχουν είναι οι επιβάτες. Δεν συμβαίνει πια αυτό. Έγινε λοιπόν μια μεγάλη αλλαγή τα τελευταία δέκα χρόνια για το πώς λειτουργούν οι φορείς των σιδηροδρόμων και νομίζω ότι όλοι συμβάλαμε ε, στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης για να γίνει αυτή η κίνηση. Άλλη λοιπόν, άλλο ένα βήμα ε, προόδου και που πρέπει να κάνουμε δηλαδή και όμως και να, προσφε... να, να πιέσουμε και άλλωστε να υπάρξει και άλλη κίνηση. Κάνετε πολλά σχόλια. Επιτρέψτε μου να τα διεξέλθω. Χρηματοδότηση πρώτα ο κ. Γκρός, ο κ. Κράμερ, ο κ. Ρικέ, η κ. Μάισνερ και άλλοι. Εάν εξετάσετε την ανακοίνωση που βάλαμε, θα δείτε ότι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τουλάχιστον, τηρούμε τις υποσχέσεις μας ότι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, δηλαδή πάνω από 60% οι σιδηρόδρομοι ε, από τα κονδύλια αυτά. Βέβαια είναι λίγα σε σχέση με τα περιφερειακά και διαφορετικά ταμεία. Περίπου 80 δις για ε, έργα μεταφορών και από αυτά περίπου 25 για σιδηροδρομικά. Παρ' όλα αυτά είναι πολλά χρήματα. Το πρόβλημα τώρα της χρήσης των κονδυλίων αυτών για την επιβολή κυρώσεων σημαίνει ότι θα επιβληθούν κυρώσεις σε ορισμένες χώρες μέλη και όχι σε άλλες. Είναι η παλιά συζήτηση αυτή. Διότι τα περιφερειακά ταμεία κάθε αυτά πάνε σε ορισμένες χώρες μέλη και όχι σε άλλες. Και αν εξετάσετε την λίστα των ενόχων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι περιλαμβάνει τους σωστούς ενόχους η λίστα αυτή. εάν δηλαδή προσπαθείτε να επιβάλλετε κυρώσεις μέσω των χρηματοδοτήσεων. Δηλαδή ορισμένοι, θα, ορισμένοι ένοχοι θα ξεφύγουν. Άρα το μόνο που μπορεί να κάνει κανένας είναι να πάει στο δικαστήριο, να εκδώσει το δικαστήριο απόφαση, να εφαρμοστεί. Εάν δεν εφαρμοστεί, να επανέλθει κανείς σε προσφυγή και τότε να μπορέσουν να επιβληθούν κυρώσεις σε όλες τις χώρες μέλη. Και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα. Είναι κάπως ιδιαίτερη κατάσταση. Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις αλλά και, και οι επιχειρήσεις που παράγουν τροχαίο υλικό αντιλαμβάνονται ότι πέρασαν, πέρασε ο χρόνος, τελείωσε ο χρόνος τους, διότι αν δεν τα καταφέρουμε τελικά καλά στην Ευρώπη όλοι θα καταλήξουμε να αγοράζουμε κινέζικα βαγόνια ή δεν ξέρω από ποιες άλλες χώρες. Διότι έχουμε κατακαιρματίσει προβολικά τις αγορές. Τελικά τα προϊόντα αυτά γίνονται ιδιαίτερα υπερβολικά ακριβά στις ευρωπαϊκές αγορές και νομίζω πάλι επιστρέφοντας στο πρόσφατο παρελθόν στον τομέα των σιδηροδρόμων η καλύτερη σύμμαχή μας για να προχωρήσουμε τα πράγματα είναι οι κατασκευαστές τροχιού υλικού αλλά και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται ότι είτε τελικά θα χάσουν και θα κερδίσουν οι άλλοι, οι άλλοι τρόποι δηλαδή μεταφορών, ή θα κερδίσουν οι άλλοι παραγωγοί. Εάν δεν τα καταφέρουμε δηλαδή πραγματικά να φτιάξουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή σιδηροδρομική αγορά που να έχει το κρίσιμο μέγεθος ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν όλες οι επιχειρήσεις και εσωτερικά στον εσωτερικό ανταγωνισμό αλλά και εξωτερικά ε, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αλλιώς δεν έχουμε άλλη δυνατότητα γιατί στο υπόλοιπο του κόσμου ε, ζουν μια αναγέννηση των σιδηροδρόμων και στις Ινδίες και στην, Κεντρική, και στην ε, Λατινική Αμερική και στη Βόρεια Αμερική και Δηλαδή έχει νόημα και από οικονομική σκοπιά αυτό. Και όσο το συντομότερο το τηληθούμε, τόσο το καλύτερο. Με την έννοια αυτή η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, δηλαδή το τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ώστε εκτός από το εύρος της τροχιάς και τα βολτ, δηλαδή το, το, το τροχαίο υλικό να μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις ε, χώρες μέλη και όχι να περνά από 5 και 6 διαδικασίες ε, διαπίστωσης της ασφαλούς λειτουργίας στις διάφορες ε, επιμέρους αγορές. Αυτό λοιπόν πρέπει επίσης να μας απασχολήσει. Βέβαια αυτό δεν εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια αναδιατύπωσης, αλλά πρέπει να μπει. Τώρα να μην αρχίσω μια ενδογερμανική συζήτηση Δεν είναι βέβαια μόνο η Γερμανία κατά της οποίας γίνεται προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουμε συνολικά πέντε χώρες μέλη. που έχουν ακόμα ελλείψεις στην οργάνωση των συνδρομικών τους επιχειρήσεων. Προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τι σημαίνει αυτό. Διαφωνήσαμε, εν τέλει τώρα θα καταλήξουμε ενώπιον του δικαστηρίου για να δοθεί σαφήνεια και ελπίζω να προκύψει σύντομα η απόφαση και ελπίζω ταυτόχρονα σε μια διετία να υπάρχει και η νομοθεσία, να εγκριθεί και η νομοθεσία, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των εγχώριων αγορών μεταφοράς επιβατών, δεν μπορεί το θέμα εδώ να είναι μόνο ο ανταγωνισμός. Γνωρίζουμε ότι στην αγορά των επιβατικών μεταφορών δεν μπορεί να διατηρηθεί η αγορά αυτή μόνο με ανταγωνισμό. Πρέπει να σκεφτεί κανείς και τις υποχρεώσεις του δημόσιου τομέα, τα κριτήρια ποιότητας, αλλά και κάποιο ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Άρα πρέπει να διασφαλίσει κανείς πολύ ευχαρίστω θα συζητήσουμε και μαζί σας τα στοιχεία που χρειάζεται να περιληφθούν, αλλά πώς μπορεί να διατηρηθεί να ε, διατηρηθούν προδιαγραφές υψηλής σα ποιότητας, ταυτόχρονα όμως να διευκολυνθεί ένα άνοιγμα των εγχωρίων αγορών. Δεν θα έλθω σε προσωπικές μου εμπειρίες, αλλά σε χώρες μέλη όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι υπηρεσίες είναι καλύτερες από εκείνες τις υπηρεσίες που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες έχουν ανταγωνισμό. Και αυτό λοιπόν πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. έδωσα κάποιες εστογενικές απαντήσεις. Υπήρχαν όμως και πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Δέχομαι την άποψη Ζαπανόφ για το θέμα του θορύβου. Βέβαια, είναι και εδώ το θέμα της εσωτερικής του εξωτερικού κόστους. Εάν ταυτόχρονα δημιουργείται ένα σύστημα επιδοτήσεων, δεν προβαίνεται τότε σε εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους, αλλά λέτε στη χώρα μέλος, έχει καλώς, επιδότησε την εφαρμογή συστημάτων τεχνολογίας ή οτιδήποτε άλλο για να μειωθεί ο θόρυβος, αλλά ο τρόπος που διατυπώνεται στην αναδιατυπωμένη πρόταση είναι ανοιχτό ακόμη. Για την οικία Τσικάου, για το e ITMS, τη συζήτηση αυτή δηλαδή. Από το 2015 και μετά στοχεύουμε στις εκπτώσεις, 5% και μετά φθήνοντας και για τις επιβατικές μεταφορές από το 2020. Και με τα σχέδια ανάπτυξης του ΙΑΤΕΜΕΣ αλλά θα έχουν ένα κάποιο πλεονέκτημα μόνο οι πρώτες οι επιχειρήσεις, δηλαδή οι πρώτες ερχόμενες επιχειρήσεις να βελτιώσουν το τροχιό του υλικό με επενδύσεις του ETMS. Ε, μη διατηρώντα έτσι ίσως όρου ανταγωνισμού. Προσπάθησα με κάπω γενικό τρόπο να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Τώρα που είμαστε σοφότεροι, κύριε Ρικέ, λέμε και εμείς ότι ίσως έπρεπε να είχαμε κάνει μόνο ένα ε, πακέτο τότε το 2000 αλλά τώρα μια και το έχουμε, α προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε το δυνατόν σύντομότερο και στα άλλα στοιχεία και σε άλλες επενδύσεις. Ε, το παιχνίδι αυτό, το the Tank Engine, κοιτάξτε εδώ χρειαζόμαστε όντως συνεργασία των, των ρυθμιστών μάλλον μεταξύ τους για να δημιουργηθεί και ένα δίκτυο συνεργασίας ρυθμιστών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δέχομαι λοιπόν την παρατήρησή σας. Πολύ από τη συζήτηση που θα γίνει και του χρόνου με την μελέτη και την νομοθετική πρόταση και όντως 75% δεν χρησιμοποιούν τα τρένα μεγάλης ταχύτητας αλλά άλλα τρένα. Θα το εξετάσουμε αυτό. Ελπίζω τέλος πάντων το περίφημο αυτό παιδικό τρένο Thomas Tetan να μπορέσει να προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα προς τα εμπρός και να μεταφέρει τους επιβάτες του όπως πρέπει. Τώρα, εύχομαι, γιατί νομίζω ότι υπάρχει πράγματι και γνήσιο το αίσθημα, είναι γνήσιο το αίσθημα της ε, βιομηχανίας ότι όντως χρειάζεται κάποια αλλαγή. Εάν αντιλαμβάνεται πράγματι η βιομηχανία αυτή την ανάγκη αλλαγής και μπορεί να ξεπεράσει ε, αυτά τα ανακλαστικά της που, που πάνε να πει δηλαδή ότι ε, της λένε τα ανακλαστικά αυτά να μείνει απ' έξω τότε αν μπορέσει λοιπόν να το ξεπεράσει αυτό τότε θα έχουμε μεγάλη πρόοδο τα επόμενα δύο χρόνια στην αγορά σιδηροδρόμων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Ρόιτε για τις απαντήσεις σας δέχομαι αυτά που λέτε για την βιομηχανία. Όντως οι σιδηρόδρομοι άλλαξαν. Αυτό ίσως μπορεί να ταρακουνήσει ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις. Εκεί βρίσκεται και το πρόβλημα. Τελειώνοντας ένα σχόλιο για τις, μετα... Ε, προμήθειες που γνωρίζετε ότι μας απασχολούν. Για τις προμήθειες τροχαίου υλικού εμείς εδώ στην Ευρώπη παίζουμε το παιχνίδι έντιμα. Ενώ στην Ιαπωνία αρνούνται να δεχθούν συμμετοχή με υποβολή προσφορών των δικών μας βιομηχανιών στην αγορά τους. Και πρέπει να το συζητήσουμε με τους Ιάπωνες αυτό. Ίσως και εμείς λοιπόν θα πρέπει να αποκλείσουμε τους Ιάπωνες από άλλες αγορές εάν συνεχίσουν να αποκλείουν τους δικούς μας κατασκευαστές από την αγορά τροχιοϊλικού σιδηροδρόμων. Εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσουμε να, εργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε μαζί σας και ίσως κάποτε να υλοποιηθεί το όνειρό μου να δω δηλαδή μια ενιαία αγορά σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά διάλειμμα.